Diamo inizio. Να ξεκινήσουμε. We start with COVID. Well, we just to... Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José Ξεκινούμε. Παρακαλώ καθίστε. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε, λέμε. Διερμηνείς με ακούτε. Συνάδελφοι, ο Επίτροπος Νταλή μας ζήτησε να αναβάλουμε την ανταλλαγή απόψεων κατά μισή ώρα, διότι είναι σε επίσημο γεύμα με την κυρία Μέρκελ. Εάν συμφωνείτε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Μποβέ. Του κυρίου Μποβέ με θέμα την αλυσίδα διανομής των ε, γεωργικών λοιπασμάτων. Δομή και συνέπειε. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και αν συμφωνείτε, κατόπιν της αλλαγής αυτής, ξεκινούμε. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 4 ε, Ιουλίου, 11-12 Ιουλίου, 30 Αυγούστου. Υπάρχουν παρατηρήσεις για αυτά τα πρακτικά. Εάν όχι, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θεωρείται εγκεκριμένο ε, εγκεκριμένα τα πρακτικά. Θα έχουμε και web streaming σήμερα στην ε, συνεδρίαση και πηγαίνουμε απευθεία στο σημείο 5 ώστε να έχει ο κύριος Νταλή το χρόνο να έρθει. Και μετά θα ξαναπάμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Πέμπτο σημείο λοιπόν, ο Νόνο είναι εδώ μαζί μα. Έκθεση του κυρίου Μποβέ για την αλυσίδα προμήθεια των γεωργικών εισρωών. Διάρθρωση και προεκτάσει. Σα θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 17 Οκτωβρίου στι 12 το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε την έκθεση στι 23, 23 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Άγκρη. Καλωσορίζουμε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στον Ζωζέ Μποβέ. Ζωζέ. Κυρίες και κύριοι, δεν θα μακρηγορήσω. Ε, θέλω απλώς να κάνω μια σύντομη παρουσίαση διότι έχουμε να κάνουμε με μια έκθεση πιστεύω ενδιαφέρουσα. Δίνει συνέχεια σε μια σειρά από εκθέσεις που επεξεργάστηκε η Επιτροπή μας και υπερψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο, όπως το ψήφισμα του Ιουνίου για την διατροφή και την ε, βιώσιμη διαχείριση των εδαφών, για την έκθεση που είχε γίνει για το ισότιμα εισοδήματα, και επίσης για το έλλειμμα των φυτικών πρωτεϊνών. Μια σειρά λοιπόν εκθέσεων που έχουν επεξεργαστεί και τα μέλη της Επιτροπής όπως ήδη από το 2008 για τη χαμηλή κατανάλωση εισρωών και σήμερα καταλήγουμε στο εξής. Μπορούμε να πούμε ότι για να έχουμε γεωργία που θα επιτρέπει ένα εισόδημα λογικό για τους γεωργούς και καλή διαχείριση των εδαφών, θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στι εισρωέ. Το ξέρετε, όπω και εγώ, ότι η κατάσταση με τι τιμέ στις διεθνεί αγορές που συνεχώ κυμαίνονται ε, χτυπά το εισόδημα των γεωργών. Το θέμα του κόστου τη παραγωγή έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε. Απλώ γνωρίζουμε σήμερα ότι το κόστο των εισρωών ε, στη Γεωργία έχει φτάσει μεταξύ του 2000 και του 2010 την αύξηση του 40% για τα γεωργικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα τελικά έχουμε αύξηση που κοστίζει πολύ ακριβά στους ίδιους τους γεωργούς. Ταυτόχρονα Αυτά τα προϊόντα ετοιμάζονται από επιχειρήσεις όλο ένα και λιγότερες. Έτσι λοιπόν έχουμε την, ε, το ρόλο των χημικών αγροτικών βιομηχανικών, αφού έξι εταιρείε μόλι ε, διαχειρίζονται το 75% τη αγορά. Ενώ μερικέ ακόμη το 45% τη αγορά. Μάλλον από αυτέ οι μεγαλύτερε το 45%. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την αγορά των γεωργικών προϊόντων και η κατάσταση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει. Δεν θα περάσω σε όλου του προβληματισμού μα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το νερό, τη διαχείριση των υδάτων, το κόστος των γεών, είτε εκμισθώνονται είτε πολλούνται, για το ζήτημα της πρόσβασης στη γη, την γεωκτημοσύνη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όλο και σημαντικότερο για τους γεωργούς. Για τις πορές μπορούμε να μιλήσουμε, για τους πόρους, για το κόστος των πράσινων μεθόδων, για το κόστος των τροφών στην κτηνοτροφία, για τα κοπάδια, ιδίως τη σόγια. Οι διακοιμάσει στι τιμέ δημιουργούν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα και εντάσει, τριγμού. Πέραν αυτών υπάρχει και μια σειρά από προτάσει τις οποίες έχω ετοιμάσει, δεν θα τις εξηγήσω κατά Θα χάσουμε πολύ χρόνο και ο καθένας τα χαρτιά του μπορεί να τα διαβάσει. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ποια θα είναι η προσέγγισή μας. Είναι να ασχοληθούμε, με να δημιουργήσουμε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πιο αυτόνομες, ανεξάρτητες και οι πρακτικές που θα ε, εξασκούν να γίνονται πιο οικονομικές. Ουσιαστικά καταλήγουμε σε προτάσεις περί ελέγχου των εισρωών, γεωπονικές προτάσεις που έρχονται να συμπλέψουν με τα όσα περιλαμβάνει ΚΑΠ και ιδίω για την ε, μετακύληση των για την άμυψη σπορά Επίσης, ε, συνεργαζόμαστε με τις δημόσιες αρχές για να βεβαιωθούμε ότι όλες αυτές οι πρακτικές μπορούν να πλαισιώνονται σωστά και να αναγνωρίζονται καλύτερα. Όλη η δουλειά αυτή λοιπόν πρέπει να γίνει στο επίπεδο τη αγρονομία και γεωπονική. Επίση το θέμα τη γεωκτημοσύνη, γιατί εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο να περιοριστεί και να αναχαιριστεί ο πληθωρισμό των τιμών τη γη. Επίση το θέμα τη ενέργεια. Ε, Ω προ την ενέργεια βλέπουμε καλά τι συμβαίνει σήμερα. Πρέπει να σταματήσουμε την κατασπατάληση της ενέργειας και να αξιοποιούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους ενεργειακούς μας πόρους στις εκμεταλλεύσεις, λόγω χάρη με πηγή τα απόβλητα, ώστε μπορέσουν οι γεωργοί να χρησιμοποιούν τα απόβλητά τους για να παράγουν ενέργεια. και αυτό στο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, <clears throat> αξιοποιώντα διαφορετικού είδου πιστώσει. Θέλησα με την έκθεση αυτή λοιπόν να παρουσιάσω όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία προτού φτάσουμε στο επίπεδο της παραγωγής και που βεβαίως επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των γεωργών. Δεν θα περάσω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Έχετε τα έγγραφα στα χέρια σας. Το σημαντικό είναι να συντονιστούμε στην εργασία μας. Αρχικά δεν υπήρχε εισηγητής για το θέμα αυτό, αλλά μετά από βραχικύκλωμα που προέκυψε σε άλλη ομάδα, ήρθε εισηγητής και από άλλη ομάδα. Με την κυρία Μαγκίνης, λοιπόν, συνεργαστήκαμε για, την, ε, για τον έλεγχο της έκθεση αυτής. Ελπίζω ότι θα ικανοποιηθεί με το περιεχόμενο της έκθεσης και την ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη της. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε, γιατί επιθυμώ η έκθεση αυτή να προχωρήσει, να φτάσει στην Ολομέλεια. Ίσως κάποιοι να θελήσουν να θέσουν και προφορικό, προφορική ερώτηση για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν είναι η καταλληλότερη στιγμή. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε μια κοινή θέση η οποία να συσχετιστεί ξεκάθαρα με το σχέδιο μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Νομίζω ότι τα ζητήματα που καλύπτει η έκθεση συσχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα αυτό. Κυρίως τα αγρονομικά ζητήματα, οι γεωπονικές πρακτικές, που θα επιτρέψουν και τον περιορισμό των εισρωών, την καλύτερη άμεψη σπορά και την ε, εξάσκησή της και βεβαίως τη βελτίωση του εισοδήματος των γεωργών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ζωζέ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση ο Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο Ζωζέ Μποβέ για το σχέδιο έκθεσης που μας υπέβαλε. Υπάρχουν αρκετά συγκλονιστικά στοιχεία ε, στην έκθεση αυτή, ό,τι αφορά την κατά 60% αύξηση στην ενέργεια και κατά 80% τη αύξηση του κόστους ε, λιπασμάτων. Η αύξηση του κόστους των ισρών είναι συγκλονιστική και μας συνταράζουν. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο κατά πόσο προτείνει στην έκθεσή του ή θα προτείνει ηλεκτρονική ταυτοποίηση των βοηδών και το επιπλέον κόστος ε, που επιβάλλει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γενετικώς ε, βελτιωμένα ε, για τις γενετικώς βελτιωμένες φυτικές ποικιλίε. Σας ευχαριστώ κύριε Νικολέσκου, κύριε Ρέμερς και μετά κύριε Μαγκίνες. Εγώ νομίζω ότι μιλώντας για τα έξοδα των εκμεταλλεύσεων πρέπει να μιλούμε και για το κόστος που επιβάλλει η κοινοτική γραφειοκρατία, ε, τα διάφορα έγγραφα, η συμπλήρωσή τους κλπ. Και έχω την εντύπωση ότι τελευταία αγνοείται η ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας και ότι εκπονούνται και ψηφίζονται και εγκρίνονται όλο και περισσότεροι κανονισμοί και διατάξεις που είναι σε βάρος των των γεωργών αυτόν τον παράγοντα κόστους με ποιον τρόπο θα τον αντιμετωπίσουμε και πώς θα τον μειώσουμε. Δεύτερο, σημειώνω ότι ιδίω στην Γερμανία, όπου βεβαίως στον τομέα της βιοενέργειας είμαστε αρκετά προχωρημένοι, βλέπουμε προώθηση της βιοενέργειας, της βιολογικής ενέργειας, όπως θέλουμε πραγματικά να γίνει, αλλά αυτό οδηγεί σε αύξηση του κόστους της γης και για την αγορά και για την ε, μίσθωση. Το ίδιο για την βελτίωση της εξέλιξης της ενιαίας αγοράς. Είναι και αυτό και, και εκεί επιβλαβές. Δηλαδή χάνονται οι γέες αυτές διότι δεν καλλιεργούνται πλέον για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τροφίμων με άλλα λόγια. ώστε τα αντισταθμιστικά μέτρα να μην αναφέρονται πάντα μόνο σε επιφάνεια αλλά και, σε άλλο, και με άλλους τρόπους και να βρεθούν άλλες ρυθμίσεις και να σκεφτούμε ακόμη εάν με διάφορα μη δασμολογικά κολλήματα οδηγούμε στο μέλλον στην αύξηση της τιμής των πόρων και για τους γεωργούς. Θα συνεχίσουμε ως Ευρώπη να παίζουμε το δικό μας ιδιαίτερο παιχνίδι ή θα προσαρμοστούμε όλο και περισσότερο στην παγκόσμια αγορά. Ευχαριστώ Μπέτα. Μαγκίνης, ευχαριστώ και εσάς και τον εισηγητή για την εισαγωγή στην έκθεσή του αλλά και για την έκθεση την ίδια. Η ιδέα στην οποία βασίστηκε η έκθεση είναι ότι τώρα που αυξάνουν οι τιμές των γεωργικών προϊόντων όλοι νομίζουν ότι τα πράγματα πάνε καλά στη γεωργία αλλά εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας πρέπει να πιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυξάνονται, αυξάνεται το κόστος των εισρώων και μάλιστα ταχύτερα από ότι αυξάνεται το κόστος των υλικών που πολλούν οι γεωργοί. Επομένως, στην έκθεση ίσως πρέπει να τονίσουμε περισσότερο, για παράδειγμα, το θέμα της τιμής της ενέργειας για τη γεωργία. Μιλούμε για την αγροτική παραγωγή της Ένωσης. Το ίδιο στον χώρο της τιμής των γεών. Και αυτό είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, παράγραφος 22. Μου φαίνεται καλή η ιδέα της δεξαγωγή μελέτης. Δεν είμαι βεβαία εάν με την ενωσιακή νομοθεσία μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμέ των γεών. Και ε, το ίδιο και την παράγραφο G στην αρχή της εκθέσεως. Αλλά σίγουρα πάντως με κάποιον τρόπο πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το κόστος της γης και περισσότερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στις τιμές των ε, λοιπασμάτων και την αγορά τους και πώς λειτουργεί. Έψαξα να βρω σχετικέ πληροφορίες. Φαίνεται πως είναι δύσκολο να ε, αποφύγουν να αγοράζουν λοιπάσματα οι γεωργοί. Πρέπει λοιπόν να το δούμε και αυτό. Θα πρέπει να, βρούμε, να δούμε πρώτα κάποιες ενδείξεις, να βρούμε κάποιες ενδείξεις σχετικά με το κόστος των ίσρων. και τι επιπτώσει έχουν. Αν έχουν αρνητικέ επιπτώσει σε όλου του τομείς ή σε ορισμένου μόνο ειδικού τομείς. Σχετικά με το κόστο των εισρώων αυτή πλήττει το εισόδημα αλλά και την βιωσιμότητα τη Ευρωπαϊκή Γεωργίας γιατί κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου οι γεωργοί, οι παραγωγοί δεν θα παράγουν πλέον εάν δεν εξασφαλίζουν επαρκέ εισόδημα. Και αν συνεχίσει αυτή η έλλειψη ισορροπία ανάμεσα στη του κόστου των εισρώων και στην τιμή των έκροων θα έχουμε πρόβλημα σχετικά με την παραγωγή τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση πρέπει να τονίσει, θέτοντας υπόψη όλων των συναδέλφων μας Ευρωβουλευτών, τα θέματα αυτά. Για την αγρονομία και τις βέλτιστες πρακτικές, ελπίζαμε οι χώρες μέλη, στη δική τους επικράτεια τουλάχιστον, να έχουν επαρκή έρευνα για το ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ μέσα στην ίδια τη χώρα. Φαίνεται όμω πω σημαίνονται προβλήματα στον τομέα αυτό. Και παλαιότερα το έχουμε θίξει και ίσω και στην παρούσα έκθεση πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπαγορεύσουμε στους γεωργούς αναγκαστικά ποιες καλλιέργειες θα πρέπει να επιλέξουν. Οι γεωργοί ας το επιλέξουν σύμφωνα με την εμπειρία τους, με το είδος των γεών που έχουν στη διάθεσή τους, ποιε είναι οι καλύτερες ε, παραγωγές να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το να επιβάλλουμε στους ε, γεωργούς το τι θα καλλιεργούν. Αλλά μιλώντας με γεωργούς ως άτομα αλλά και ως επιχειρηματίες διαπιστώνω ότι ανησυχούν πολύ για την αύξηση του κόστους των ισρών. Τέλος, παράγραφος 4 κύριε Πρόεδρε που μιλεί για νομοθεσία antitrust. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν και μάλιστα και πρόσφατα πέρσι μόνο έχουν επιβάλει πρόστιμα σε ορισμένες ε, επιχειρήσεις γιατί είχαν συμπήξει καρτέλ. Ίσως λοιπόν έχουμε επαρκή νομοθεσία για την ώρα, έτσι θεωρώ. Το ζήτημα είναι η συλλογή και παροχή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, ότι δηλαδή η συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών είναι αντιανταγωνιστική. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και προσεκτικοί στι διατυπώσει που θα επιλέξουμε. Έχουμε πάντω χρόνο για να καταθέσουμε και να συζητήσουμε τροπολογίε και αναμένω από τον εισηγητή να, να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρέιντ. Ο κύριος Τογιανόφ και μετά ο κύριος Καπολάς Σάντους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό που η Επιτροπή μας ασχολείται με το θέμα αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που την έκθεση αυτή την ανέλαβε ο κύριος Μποβέ γιατί νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος ε, για την κατάλληλη έκθεση. Σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα που διατύπωσαν οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλονται σε μεγάλο βαθμό από τι δράσει μα και την πολιτική μα του παρελθόντο. Ο κύριος Νικολέσκου είπε κάτι παρόμοιο και η αύξηση των τιμών παραγωγής ήταν κάτι που συζητήσαμε επί μακρόν. Αλλά τώρα έχουμε ακόμη πιο αυστηρές απαιτήσει στην παραγωγή μας. Για μία εξαετία ήμουν αρχικά παρατηρητής, μετά έγινα ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και άλλων επιτροπών. Και πιστεύω ότι η γεωργία είναι ο κλάδος που πλήττεται το επιτοπλίστων. Είναι πολύ πιο αυστηρή η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στη γεωργία από ό,τι απέναντι σε άλλους ε, κλάδους της οικονομίας. Και αυτές οι υψηλές απαιτήσει αυξάνουν και το κόστος. Επιπλέον ε, εντείνεται το γραφειοκρατικό άχθος, όπως ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι, και αυτό επιβαρύνει τους γεωργούς. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιήσουμε, λέμε, τους γεωργούς, αλλά χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση, καλύτερες, περισσότερες εξηγήσει και δυστυχώ δεν λαμβάνουν αυτή τη συμπληρωματική πληροφόρηση για να ανταπεξέλθουν στι υποχρεώσεις που του απαιτούνται. Επίση, ε, παρατηρούμε ένα σχεδόν μονοπόλιο στα διάφορα υλικά των ισρώων. Η Βουλγαρία είναι κατά παράδοση αγροτική χώρα και είχαμε ένα είδο ε, ε, αυτάρκειας στη Γεωργία που δυστυχώς έχει εξαλειφθεί και μάλιστα εξαλείφθηκε σχεδόν από την μέρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην Βουλγαρία, στο παρελθόν είχαμε ε, μεγάλα εργοστάσια παρασκευής τέτοιων χημικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων, αλλά μετά από πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασαν τα εργοστάσια αυτά σε ε, ιδιώτες. Και τώρα δημιουργήθηκε ένα de facto μονοπόλιο στην αγορά, όπως επισήμανε και ο κύριος ε, ε, Μποβέ. Αρχικά τα εργοστάσια αυτά ήταν μικρά σε σχέση με τις διαστάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα μικρά εργοστάσια εξολοθρεύθηκαν και μάλιστα θεωρώ ότι έγινε σκεμμένα αυτή η εξολόθρευση προκειμένου να ευνοηθούν τα μονοπόλια και αυτή η συγκέντρωση που ακούσαμε. Οπότε δημιουργήθηκαν κάποια μονοπόλια, συνήθισαν συμφωνίες καρτέλ και συγκέντρωσης και το ίδιο ισχύει και για μερικά Ινστιτούτα, γεωργίας, οι οργανώσεις που αρχικά παρήγαγαν συγκεκριμένα είδη σπόρων ή συγκεκριμένα γονίδια για τις ζωοτροφές. Και όλα αυτά καταστράφηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα η χρηματοδότηση τέτοιων ερευνητικών ε, γεωργικών κέντρων, η χρηματοδότηση έχει μειωθεί, οπότε και τα νέα αυτά ερευνητικά κέντρα δεν παράγουν νέα προϊόντα. Υπάρχει και ένα στοιχείο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ε, λεγόμενη πράσινη ενέργεια. Και διαπιστώνουμε ότι είναι υψηλό το κόστος της ενέργειας, αλλά δεν νομίζω ότι η εκτίμηση της έκθεσης είναι σωστή. Σίγουρα η πράσινη, η πράσινη ενέργεια μας ενδιαφέρει και θέλουμε να την αναπτύξουμε, αλλά η σημερινή κατάσταση και η πολιτική μας οδηγεί σε αύξηση των τιμών καταναλωτή που έχει άμεσο αντίκτυπο στους τομείς που χρησιμοποιούν εντατικά την ενέργεια, όπως είναι η γεωργία. Ωραία όλα αυτά που λέμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε τους Αγιοργούς, αλλά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο. Και το ίδιο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργεια χρησιμοποιεί γεωργικέ ε, γέε για την παραγωγή τη. Και αυτό μειώνει τι εκτάσει εκτάσεις των καλλιεργήσιμων ε, εδαφών και ταυτόχρονα αυξάνει το τίμημα στη μίσθωση των γεών. Το αντιμετωπίζουμε αυτό στη Βουλγαρία. Ε, για τέτοιου συμβάσει απαιτείται τουλάχιστον τετραετία, τετραετή διάρκεια έως συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αντίθετα, αν κανείς μισθώσει διαμέρισμα θα πρέπει να έχει περιορισμένο χρόνο. Ενώ αν, αν μισθώνει η γη μπορεί να την εκμισθώσει επαορίστου. Κάτι που δημιουργεί πρόσφορα έδαφος για απάτες. Επίσης έτσι δημιουργούνται τεράστιες ε, γεωρικές εκμεταλλεύσεις και αποφελούνται έτσι οι μεγαλοκαλλιεργητές από τις άμεσες πληρωμές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και εμπόδια στους μικροκαλλιεργητές να χρησιμοποιήσουν τα κοινοτικά προγράμματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Στογιάννοφ, ο κύριος Καπόλα Σάντος και μετά ο Τζορτζ Λάιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω και προσωπικά, αλλά να αναπληρώσω και τον κύριο Σπύρο Δανέλη, που είναι ο σκιώδης ηγητής Σοσιαλιστικής Ομάδας και δυστυχώς απουσιάζει σήμερα. Θα ήθελα να εκφράσω στον εισηγητή μας την ικανοποίησή μου για την έκθεσή του που είναι μια καταπληκτική βάση εργασίας για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αναφέρεται ότι στην τελευταία δεκαετία το, κόστος, το ενεργειακό κόστο αυξήθηκε κατά 60%. Το κόστος λιπασμάτων αυξήθηκε κατά 80%. Ε, για τις μηχανήματα 30%, για τους σπόρους 30%. Ενώ η αύξηση των, της τιμής γεωργικών προϊόντων ήταν ε, μισή σε σχέση με τις αυξήσεις των τιμών ισρών. Κάτι που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για τους γεωργούς. Είναι ισορροπημένος ο τρόπος ε, που προσεγγίζει το πρόβλημα ο εισηγητή και τι διάφορε πτυχέ του προβλήματο, γιατί είναι πολύ σύνθετο. Γι' αυτό και θα τον υποστηρίξουμε. Παραλαμβάνω, η έκθεση είναι μια θαυμάσια βάση εργασία και θα τη βελτιώσουμε με τι τροπολογίε μα. Γιατί αυτό είναι και ένα καλό τρόπο για να ασκήσουμε κάποια επιρροή στη συζήτηση, στις συζητήσεις που θα γίνουν για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Υπάρχει μια παράληψη, κύριε Μποβέ. Πολύ σωστά και αρκετά μιλάτε για το νερό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως τις γνωστές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι προτάσεις που το περιεχόμενο του είναι γνωστό αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί επίσημα. Από ό,τι έμαθα πάντω, διαπιστώνεται ότι στο πακέτο για την ανάπτυξη τη υπαίθρου αποκλείεται από την επιλεξιμότητα το θέμα των επενδύσεων σε αρδευτικά συστήματα ενώ σε ορισμένες χώρες το θέμα της άρδευσης είναι σημαντικό και το να αποκλειστεί η επενδύση στην άρδευση από το πακέτο της Επιτροπής είναι πραγματικά συμβίβαστο και παράδειγμα. Χθε είχαμε στην Πορτογαλία θερμοκρασία 36 βαθμών Κελσίου και οι παραλίες ήταν κατάμεστες. Είχαμε αντίστοιχο θέαμα με αυτό του Αυγούστου. Αυτό λόγω των κλιματικών αλλαγών. Και στι χώρε του Νότου, χωρί ε, αποτελεσματικά συστήματα άρδευση, είναι αδύνατον να έχουμε ανταγωνιστική γεωργία. Αυτό το σημείο λοιπόν θα πρέπει να υπογραμμιστεί περαιτέρω και να βελτιωθεί στην έκθεση. Πάντως σε γενικέ γραμμέ, όπω είπα η έκθεσή σα μα βρίσκει σύμφωνος, μα ικανοποιεί μας ικανοποιεί. Συγχαρητήρια για την πυγμή σα και για την ισορροπημένη σα έκθεση. Ευχαριστούμε Λουίς. Ο κύριο Τζορτζ Λάιν και μετά Αγνιού. Πρόεδρε, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Ζωζέ Μποβέ για την έκθεσή του. Νομίζω ότι πράγματι μας δίνει καλό υλικό για να προχωρήσουμε. Δεν συμφωνώ φυσικά με όλα όσα περιέχει η έκθεση. Όμως ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια κοινή αντίληψη για τα περισσότερα ζητήματα. Τονίζει τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γεωργοί, οι οποίοι πιέζονται. Μεταξύ λίγων πολυεθνικών που είναι οι βασικοί παρέχοντες και από τις τιμές ε, στο άλλο άκρο της αλυσίδα που είναι η λιανική πώληση. Είναι πολύ δύσκολο ένας μικρός εμπορευόμενος να έχει το ανάστημα και την πυγμή για να αντισταθεί στις πιέσεις που ασκούν οι πολυεθνικές με δεσπόδουσες θέσεις και ως πολιτές των εισρώων και αγοραστές των προϊόντων που ετοιμάζουν οι γεωργοί. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε είναι με τι τρόπους θα ενισχύσουμε το ρόλο των γεωργών. Βλέπουμε ότι το κίνημα των συνεταιρισμών είναι ήδη κάτι που προχωρά και αναπτύσσεται και για την λιανική πώληση, αλλά ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε ανάλογες κινήσεις και για τις εισρωές προς τις εκμεταλλεύσεις. Ίσως οι γεωργοί από κοινού να θέλουν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά για να εμπορευτούν τα προϊόντα που παράγουν. Κάτι ακόμη που θέλω να θίξω είναι το κόστος των ζωοτροφών για τους παραγωγούς βόλου, πουλερικών και χοιρινού. Η εισαγωγή σόγιας, βασικό συστατικό για οποιαδήποτε στάδιο της κτηνοτροφίας, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα η τιμή της όγια βαρύνει τους γεωργούς αυτούς, να τα αναγνωρίσουμε. Και η Μαρέντ σωστά είπε στη συμβολή της ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την βιομηχανία λιπασμάτων. Όταν ασχολήθηκα εγώ ίδιος με τις καλλιέργειες, ε, το δυσκολότερο ήταν η τιμή των λιπασμάτων, ακόμα και μέσω των συνεταιριστικών ε, οργανισμών μας. Από έναν βασικό παραγωγό λιπασμάτων και χημικών έπρεπε να προμηθευτούμε το υλικό και είναι και βασική η εταιρεία σε όλη την Ευρώπη αυτή. Οι εταιρείε λοιπόν που είναι αυτέ που φτιάχνουν τα λοιπάσματα δεν μπορεί να παρακαθούν με τίποτα. Και όσο και αν έχουμε απευθυνθεί σε αρμόδιε αρχέ, όσο και αν προσπαθήσαμε να προσφύγουμε στι αρχέ του ανταγωνισμού, δεν καταφέραμε τίποτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Τι να κάνουν λοιπόν οι γεωργοί όταν ζητούν τιμές για τα λοιπάσματα από δύο-τρεις εταιρείες και τελικά δεν μπορούν να τις καλύψουν. Αυτό μου φαίνεται παράδεκτο. Πώ είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρχέ ανταγωνισμού να μην ερευνούν το θέμα, να μην φτάνουν στη ρίζα του προβλήματο. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Το, τα λοιπάσματα είναι ένα από τα βασικότερα, το βασικότερο κόστος που έχουν να απομισθούν οι γεωργοί. Και γιατί ακριβώς είναι τόσο λίγη παραγωγή για να ασκούν έλεγχο στην αγορά. Η αγορά λοιπόν λιπασμάτων θα πρέπει να ελεγχθεί από τις αρχές ανταγωνισμού. Πρέπει να εξασκηθούν όλες οι αρμοδιότητε που οι αυτέ και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστούμε ο κύριος Αγνιό. Ευχαριστώ. Ζωζέ, φαντάζεσαι ότι δεν θα σε συγχαρώ. Θα είμαι όμως ευγενής. Ανησυχώ Ανησυχώ για αυτά που λες για τους σπόρους. Είναι πολύ απλουστευτικό να λες. Και απλοϊκό να λες τους γεωργούς και την Επιτροπή ότι πρέπει κανείς να αποθηκεύει σπόρους για να μην πληρώνει τους τόκους και να γλιτώνει ένα μέρος του κόστους. Ξέρουμε όμως τι πηγή εισοδήματος είναι αυτή η τόκη ακριβώς, η διαφορά στην εμπή. Κάποιοι 15 χρόνια έχουν εκμεταλλευτεί αυτή την πηγή εισοδήματο. Νομίζω λοιπόν αυτό που θέλεις να πεις είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα έπρεπε να υπάρχει η επιβολή αυτού του δασμού. Όμως δεν μπορεί να διατηρηθεί το σύστημα για πολύ καιρό εάν οι ποικιλίε δεν πληρώνονται και ακριβότερα. Γιατί ακριβώς αυτοί που εμπορεύονται τις ποικιλίε χωρίς εισόδημα δεν θα μπορούν να τις προωθήσουν στην αγορά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση για το κόστος ε, δεν νομίζω ότι μπορεί η Επιτροπή να με βοηθήσει να κλειτώσω το κόστος. Για τα πουλερικά μου χρησιμοποίησα ξεχωριστό σύμβουλο, για τις 43 εκτάσεις άλλων και ούτω καθεξής. Έτσι μπόρεσε να εξοικονομήσω στο κόστος. Γιατί ε, το κόστος όμως είναι τόσο υπερβολικό. Τι χρειάστηκε να κάνω για να αντιμετωπίσω τον υπερβολικό κόστος της αγοράς. Σκέφτηκα πώς να διαχειριστώ λόγω χάρη το κτίριο. Ε, το, η Επιτροπή μου επέβαλε τον ε, ατομική, εξατομικευμένη, τον εξατομικευμένο εντοπισμό των προβάτων. Πολύ ακριβό, λόγου χάρη. Ξέρω ότι δυσκολεύεσαι και σε ενοχλεί που με ακούς, αλλά μου επέβαλαν όλους αυτούς τους ελέγχους για τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα. Και πολλά από τα προϊόντα μου έπρεπε να αποσυρθούν από την αγορά. Οι έλεγχοι λοιπόν ακριβένουν ακόμη περισσότερο. Μην μπλέκει στην Επιτροπή λοιπόν άλλο. Αυτό πρέπει να λυθεί σε επίπεδο του ίδιου του βιομηχανικού κλάδου. Ευχαριστούμε κύριε Αγνιό. Ο κύριος Νταντάν και μετά ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το έγγραφο που εκπώνησε. Όντως είναι καλή βάση εργασίας. Με μερικά σημεία συμφωνούμε, με άλλα Δεν συμφωνούμε απόλυτα. Θα χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις. Πάντως ήθελα να υπενθυμίσω ότι αν η Ευρωπαϊκή Γεωργία ε, είχε τα τελευταία χρόνια αύξηση παραγωγής είναι ακριβώς επειδή ε, προσέφηκε σε αυτές τις ροές. Και μερικές φορές, αν δεν είναι καλά ενημερωμένοι, οι γεωργοί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τον καταλληλέτερο ή το σωστότερο τρόπο της ροές. Και αν δεν το έκαναν αυτό, όπως αναφέρθηκε, είναι γιατί το βάρος των ε, εταιριών ε, που παράγουν ήταν πολύ μεγάλο και είναι κάτι που δεν αναφέρθηκε και θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όλο και πιο συχνά βρίσκεται σε μία μέγενη ο Γιώργος. Βρίσκεται σε έναν ασφυκτικό κλειό γιατί είναι τα ίδια κεφάλαια ε, που τους ε, παρέχουν τις πρωτεσίλες και που αγοράζουν ε, τα προϊόντα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Το κεφάλαιο βρίσκεται στα ίδια χέρια, οπότε το περιθώριο του γεωργού, ουσιαστικά το περιθώριο κέρδους του γεωργού καθορίζεται από τρίτους. Και όταν ε, διαπιστώνουμε με τη ζήλο η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προσπαθεί να εμποδίσει τους γεωργούς να συσπηρωθούν σε ευρύτερο όργανα από ότι συνεταιρισμούς ή οργανώσεις παραγωγών. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στα απορροκυπευτικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε για το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού στον γεωργικό κλάδο. Και νομίζω ότι σε σχέση με αυτό που θα κληθούμε να πραγματοποιήσουμε για το μέλλον της ΚΑΠ και αυτό το σημείο καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Μισελ Νταντά. Να καλωσορίσουμε τον Επίτροπο Τζον Τάλι. Μια και έχουν απομείνει μόνο τρεις ε, παρεμβάσεις, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και μετά να περάσουμε στην ανταλλαγή απόψε με τον Επίτροπο. Ο κύριος Ζωή Νίκολσον, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Ζωζέ Μποβέ για την έκθεσή του. Σίγουρα και εγώ δεν συμφωνώ με όλα που λέει, αλλά τον συγχαίρω γιατί αν μη τι άλλο μας έδωσε τροφή για σκέψη και έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Ανέφερε πολλά σημαντικά προβλήματα. Και φυσικά υπογράμμισε κάτι που όλοι γνωρίζουμε τα, τα, τα καύσιμα, τα φυτοφάρμακα και τη γη ε, τους λόγους που μερικές φορές οδηγούν σε χρεοκοπία τους γεωργούς γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν με ανταγωνιστικό τρόπο το έργο τους και οι μικροί εξολοθρεύονται προς όφελος των μεγάλων. Και με τα πουλερικά έχουμε προβλήματα στην πτυνοτροφία, για παράδειγμα, γιατί η πτυνοτρόφη εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό από τι εισαγόμενε ζωοτροφέ και οι ζωοτροφέ πραγματικά είναι σημαντικό σημείο τη εξίσωση. Και η, η και οι γενετικώ τροποποιημένε πορέ εισάγονται, κάτι που αυξάνει το κόστο των ισρώων. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ε, στο μέλλον, αλλά θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ με πολλές από τις παρατηρήσεις, γι' αυτό θα ήθελα να αποφύγω τις επαναλήψεις. Πάντως θα πρέπει να δούμε από πού συσσωρεύτηκε όλη αυτή η γραφειοκρατία. Πώς δημιουργήθηκε. Γιατί φαίνεται ότι να θέλουμε να προσέψουμε τα πράγματα, ε, εντείνουμε τη γραφειοκρατία, την ενισχύουμε. Σκεφτείτε τι άχθος θα δημιουργηθεί στις αγροτικές κοινότητες, στους γεωργούς θα εξεγερθούν με τέτοια πίεση από την γραφειοκρατία, γιατί πραγματικά το κακό έχει παρατραβήξει. Αναφέρθηκαν ορισμένα θέματα ε, και πολύ σωστά επισημάθηκαν. Υπάρχουν ε, πολλά πράγματα που επιδέχονται βελτιώσεις. Η Μαρία αναφέρθηκε και στο θέμα της γης. Και αυτό το θέμα είναι επίμαχο. Σε μια σύγχρονη κοινωνία η αξία της γης είναι αυτή που ο καθένας είναι έτοιμος να καταβάλει για τη συγκεκριμένη γη. Υπάρχουν πολλοί κερδοσκόποι, εργολάβοι, αγοράζουν οικόπεδα, αλλά αυτή η κατάσταση σχεδόν έχει εξαφανιστεί πια. Και δεν έχουμε παρόλα αυτά μείωση της τιμής της γης. Και αν δούμε όλα τα σημεία της Ευρώπης, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην αξία της γης. Πάντως, η γη σπανίζει όλο και περισσότερο και σίγουρα δεν μειώνεται η τιμή τη. Υπάρχει όλο και λιγότερη γη, όλο και λιγότερε εκτάσει, όλο και λιγότερη δυνατότητα παραγωγή. Πρέπει να αντιληφθούμε όλα αυτά τα στοιχεία, αλλιώ δεν πρόκειται να βελτιώσουμε την κατάσταση. Προσοχή λοιπόν, σπάνιο αγαθό γη, να τη χρησιμοποιήσουμε, να την αξιοποιήσουμε σωστά. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αυτέ ήταν οι απόψει μου. Ευχαριστώ και θα παρακολουθήσω με ενδιαφέρον τη συνέχεια τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ, Τζιμ. Έχω ε, συμπεριλάβει στον κατάλογο και την ε, κυρία Ράνς Καρσία. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να δευτερολογήσει στο τέλος και ο κύριος Μποβέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μποβέ γιατί πάντα είναι άξιο συγχαρητήρια για τις προσπάθειές τους και πραγματικά τα στοιχεία που μας δείχνει είναι συγκλονιστικά. Αυξήθηκαν οι τιμές των λοιπασμάτων και των συνθετικών ε, φυτοφαρμάκων κατά 80%. Οπότε προβληματίζομαι. Αν κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις πολιτικές μας αποφάσεις, όταν περιορίζουμε τον αριθμό των προϊόντων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μερικές φορές υποχρεώνουμε ή διευκολύνουμε τη χημική βιομηχανία να αξιοποιήσει ε, τις αποφάσεις αυτές και να δημιουργήσει τεράστιο κέρδος και ταυτόχρονα κάνουμε το χαζό μερικές φορές, εθελοτυφλούμε, όταν σε σημαντικές περιοχές όπως τη Μεσόγειο υποχρεώνουμε τους παραγωγούς μας να καταβάλουν τεράστιες και άδικες τιμές για τα ελληπάσματα, ενώ στην ίδια φυσική περιοχή, ε, στην νότια πλευρά της Μεσογείου, στην Βόρεια Αφρική, δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσει για τη χρήση συγκεκριμένων ε, φυτοφαρμάκων. Έχει μειωθεί κατά 15% η παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μόνο και μόνο από αποφάσει που λάβαμε αμή τι άλλο βεβαιασμένα, εσπευσμένα και σίγουρα άδικα γιατί η κατάσταση δεν είναι ίση, ισότιμη για όλους. Αναφερθήκατε σε μία ε, αρχή επίβλεψη των τιμών. Το ζητήσαμε και για την ε, αλυσίδα τροφίμων. Ζητήσαμε ένα παρατηρητήριο των τιμών. Είναι μια ακόμη απόπειρα. Θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε και σίγουρα δεν θα σταθούμε εμεί εμπόδιο στην αύξηση τη διαφάνεια. Το αντίθετο. Την επιζητούμε. Σε ό,τι αφορά την τήρηση πρακτικών φιλικών προ το περιβάλλον ή που θα σέβονται το περιβάλλον, φυσικά συμφωνώ όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και εγώ και στη ζωή είμαι υπέρ του περιβάλλοντος. Δεν βλέπω ε, κα, δεν καταλαβαίνω καλά την διάκριση που κάνετε γιατί λέτε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν θα πρέπει να έρθουν σε ανταγωνισμό με την παραγωγή τροφίμων. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι βάσιμη αυτή η ανησυχία. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι η αντίφαση που υπάρχει, που διαπιστώνω εγώ τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να συμβάσετε την αύξηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων με την μείωση των τιμών ισορών. Με την αύξηση του περιβαλλοντικού κόστου θα αυξηθεί και το κόστος των ισορών. Πώς είναι δυνατόν ε, με, τη, με τα χρήματα της ΚΑΠ να έχουν περισσότερα κονδύλια για το ε, πρασίνισμα. Εγώ βλέπω περικοπές κατά 10% των σχετικών κονδυλίων. Οπότε αν είμαστε πολύ απαιτητικοί, υπερβολικά ιδιότροποι, με την αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ε, απαιτήσεων προς τους γεωργούς θα τους υποχρεώσουμε να αναλάβουν και το κόστος, να υπομισθούν αυτή την ευθύνη και να χάσουν σε αποδοτικότητα ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τις, τους πόρους. Βλέπω ότι έχετε μια έμεση επίθεση, διαφωνία με τις γενετικώς τροποποιημένες ε, σπορές. Εγώ και ως Ισπανίδα, αλλά και προσωπικά, διαφωνώ με τη γνώμη σας και τη θέση σας για τους σπόρους γενετικώς τροποποιημένους. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, Ζωζέ, μήπω θε να προσθέσει τίποτα για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ιδάλω, πάμε απευθεία στο 4. Επιστρέφουμε δηλαδή στο 4, εφόσον έχει έρθει ο κύριο Νταλή. Ένα λεπτό, Ζωζέ. Ένα λεπτό μόνο για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Πολλά αναφέρθηκαν. Ίσως κάτι να επισημάνω στην κυρία Ράιμερ και τις, τους άλλους συναδέλφους που σχολίασαν την τιμή της γης. Να ξέρετε ότι σήμερα εξαιτία των εργοστασίων βιοαερίου των βιομηχανικών ε, δηλαδή εργοστασίων. Έχουμε φτάσει σε τιμές εκταρίων 2.000 ε, ευρώ. Φαίνεται απίθανο και απίστευτο, αλλά μιλάμε για εδάφη που τα έχουν ε, αρπάξει ουσιαστικά οι μεγάλες βιομηχανίες, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αφοσιωμένα, να χρησιμοποιούνται για την ε, καλλιέργεια τροφίμων και την παραγωγή τροφίμων. Έτσι λοιπόν, η σπορά δεν είναι κάτι καινούριο. Αναφέρεται και στην έκθεση του κυρίου Ντες. Έχουμε έκθεση λοιπόν του Κοινοβουλίου που λέει πώς οι γεωργικές πρακτικές σήμερα πρέπει να λάβουν ένα νέο προσανατολισμό. Πρέπει να περιορίσουμε λοιπόν τις εισρωές, όχι απλώς για την ευχαρίστηση, την απλή του περιορισμού, αλλά γιατί ακριβώς οι σημερινές γεωργικές πρακτικές θα μας επιτρέψουν να έχουμε χρήση, την αποθήκευση του αζώτου στο ίδιο το έδαφος και να μην έχουμε συνεχή χρήση αζωτούχων λοιπασμάτων. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και ευχαριστώ και εσάς συνάδελφοι για την πολύ συμπαθητική σας παρέμβαση. Κύριε Αγνιό, ευχαριστώ Ζωζέ. Σου δίνουμε λοιπόν τις ευχές μας για την καλή συνέχιση τη συζήτηση και του θέματο αυτού. Σημείο 4 τώρα. Καλωσορίζω τον Επίτροπο Νταλή, υπεύθυνο για την υγεία και τους καταναλωτές. Θα μας παρουσιάσει την κατάσταση και το πώς έχει προχωρήσει η οδηγία 1999-74 ΕΚ για τις και όρνηθες. Όπως τα ξέρετε, η οδηγία αυτή προβλέπει την απαγόρευση της ε, εκτροφής οτόκων ορνηθών σε συμβατικούς κλοβούς τις λεγόμενες μη διαμορφωμένου τους λεγόμενους μη διαμορφωμένους και αυτό από την 1η Ιανουαρίου 2012. Σας θυμίζω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2010 όπου το Κοινοβούλιο εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για το σημαντικό αριθμό κατών μελών και παραγωγών αυγών που δεν έχουν σεβαστεί εγκαίρως την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2012. Πέραν του θέματος των οτόκων ορνηθών, θα μας ενημερώσει ο Επίτροπος και για τις επιπτώσεις ε, από την απόφαση του δικαστηρίου για την γύρη όπου υπάρχουν ίχνη από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς στο μέλι. Κύριε Πέτρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, θα ρίξω το βάρος ιδιαίτερα σε δύο θέματα σήμερα που ενδιαφέρον την Επιτροπή, τις ΟΟΤΟ και και το θέμα επίσης της γύρης και του μελιού. Σε λίγο θα έχουμε 1η Ιανουαρίου 2012 που αρχίζει η απαγόρευση της χρήσης συστοιχειών κλοβών ορνήθων που έχει συμφωνηθεί ήδη από το 1999. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάθε ευκαιρία υπενθύμησε στις χώρες μέλη τις υποχρώσεις που έχουν αναλάβει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, σχετικής νομοθεσίας. Τον Δεκέμβριο του 2010 ε, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που στηρίζει την εφαρμογή της απαγόρευσης χωρίς καθυστέρηση και που ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της και συμμόρφωση ε, με την νομοθεσία. Τον Ιανουάριο φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε συνεδρίαση με πολλούς από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ε, απαγόρευση των συστοιχιών κλωβών ορνήθων για να καθορίσουν μάλλον το Φεβρουάριο ζήτησα από τους υπουργούς να στείλουν στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές τα αριθμητικά δεδομένα μέχρι 1η Απριλίου δηλαδή των αριθμών των ορνήθων ανακατηγορία μέχρι τον Απρίλιο. Από τα δεδομένα αυτά ορισμένες χώρες μέλη φαίνεται ότι θα εξακολουθούν να ε, διατηρούν όρνηθες σε κλωβούς μέχρι τον μέχρι τέλου του έτους. Η κατάσταση λοιπόν σε ορισμένες χώρες μέλη και πολλών ευρωπαϊκών παραγωγών η κατάστασή τους είναι άγνωστη στις αρμόδιες αρχές. Αυτό είναι σαφώς απαράδεκτο. Μετά από πολλού μήνες εντατική εργασία, εμφανίζομαι ενώπιόν σας για να επιβεβαιώσω και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να αναβάλει την ε, ημερομηνία ενάξεως εφαρμογής της απαγόρευσης και ότι θα λάβει ε, μέτρα σύμφωνα με τις ε, αρμοδιότητες που της ε, χορηγεί συνθήκη. Διότι δεν επιτρέπεται να υπονομευθούν ούτε η παραγωγή ούτε η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Θα πρέπει να, να αποφευχθούν οποιασδήποτε στρεβλώσεις της αγοράς μετά από τον Ιανουάριο 2012 είναι περιορισμένοι οι πόροι των επιθεωρήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω θα διατεθούν όλοι ω προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν, από 1η Πρώτου 2012, οι εμπειρογνώμονε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσουν να επισκέπτονται κατ' επιλογή χώρε μέλη. Και μετά από του ελέγχου αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα διστάσει να ξεκινήσει όπου αυτό είναι απαραίτητο ε, διαδικασίες επί παραβιάση μέσα στο 2012. Επίσης στο Αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών θα υπενθυμίσω αυτό τον μήνα στις χώρες μέλη τις ευθύνε τους και θα απευθύνω έκκληση σε όλους τους αρμόδιους υπουργού να το θεωρήσουν δική τους αυστηρά προσωπική προτεραιότητα να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την απαγόρευση της χρήσης των κλοβών αυτών όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στρέφομαι τώρα στους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα θέματα του μελιού. που είναι το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα λόγω δύο πρόσφατων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχουν ε, ελκύσει την προσοχή και που για το μέλη στις 6 Σεπτεμβρίου το δικαστήριο έκρινε ότι ακόμα και μικρά ίχνη γύρις από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς χρειάζονται την απαραίτητη επισήμανση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τις συνέπειες της απόφασης αυτής που είναι δύο ειδών. Πρώτον, για την παραγωγή του μελιού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο, για τις εισαγωγές μελιού από τρίτες χώρες. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνύπαρξη μεταξύ κυψελών και ε, τροποποιημένων οργανισμών είναι αυτή που προκαλεί τα προβλήματα και που δείχνει την σημασία που έχει ο έλεγχο από πλευρά χωρών μελών τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και βεβαίω ο τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση στο επίπεδο των κρατών μελών του δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τι τεχνικέ αυτέ πηχέ στις 22 Σεπτεμβρίου μαζί με τις χώρες μέλη και μίλησε και με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με την βιομηχανία τροφίμων, γεωργούς, οργανώσεις των γεωργών καθώς και των μελισσοκόμων τις τελευταίες εβδομάδες. Θα συνεχίσουμε να ερευνούμε το θέμα αυτό μαζί με το κοινό κέντρο ερευνών το οποίο αναλύει τα σχετικά θέματα. Ελπίζω δε ότι όλες οι χώρες μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αντιδράσουν με τρόπο συντονισμένο. Δεν επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατικό ή τοπικό. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, 50% περίπου του μελιού που καταναλώνουμε εισάγεται από τρίτες χώρες, όπως την Αργεντινή, την Κίνα ή τη Βραζιλία, όπου γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, εσοδίες, καμιά φορά που απαγορεύεται η χρήση τους και η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί χρησιμοποιούνται ωστόσο ευρέως. Πρόσφατα, στις 20 Σεπτεμβρίου, συζητήσαμε με τις εκπροσώπους των χωρών αυτών για να συζητήσουμε την απόφαση. Και συζητούμε ορισμένες ε, πτυχές της ρυθμιστικής νομοθεσίας για να εφαρμόσουμε τη σχετική απόφαση. Και ιδίως για την χρήση καλαμποκιού και για χρήση ορισμένων ε, ειδών τροφίμων που δεν περιέχουν γύρι. Και κάνουμε τώρα μέτρα, λαμβάνουμε τώρα μέτρα για να κλείσουμε το σχετικό κενό, δίνοντας μια έγκριση που θα καλύπτει όλες τις χρήσεις τροφίμων. Το 810 είναι γενικά, γενικά τροποποιημένος οργανισμός ο οποίος έχει εγκριθεί εδώ και μία δεκαετία. Χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις διατροφής και ε, κρίνεται ασφαλής. Ζητήθηκε από την ΕΦΣΑ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, να υποβάλει γνωμοδότηση για το καλαμπόκι αυτό και για το μέλι. Η δεύτερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι για την χρήση του καλαμποκιού το 801 από πλευράς γαλλικών αρχών. Η, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να κρίνουν την νομιμότητα των μέτρων. Επομένως, το Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας θα συναγάγει τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την ε, νομιμότητα της απαγόρευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τις επιπτώσεις της σχετικής αποφάσεως, εφόσον υπάρξει, των γαλλικών δηλαδή μέτρων διαφυλάξεως για τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο 2010 υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την καλλιέργεια των γάμα τάφων η οποία πρόταση καλύπτει το θέμα των εθνικών απαγορεύσεων ε, καλλιέργειας γαματαφόμικρων και ζητά από και κρίνει μάλλον την ευκαμψία των χωρών μελών, των ευελιξίων χωρών μελών να χρησιμοποιήσουν ε, σε καλλιέργειες τέτοιους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Χαιρόμαστε πάντως για την ταχεία αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την πρώτη ανάγνωσή σας στις 5 Ιουλίου και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει μια κοινή θέση σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Νταλή, για αυτή την ε, ενημέρωση. Και τώρα ξεκινούμε μια συζήτηση ιδιαίτερα εντατική. Όλοι οι βουλευτές που είναι παρόντες στην αίθουσα έχουν ζητήσει το λόγο. Σχεδόν όλοι, τέλος παντών και όλες. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να συγκρατηθούμε στο χρόνο ομιλίας μας, γιατί μετά θα πρέπει να μας αφήσει ο Επίτροπος. Η κυρία Γέγκλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, αν και βέβαια για τα θέματα αυτά μπορεί κανείς ε, να μιλήσει διαμακρών. Για την προστασία τώρα των οτόκων ορνήθων. Αυτό είπατε, σωστά το είπατε. Προστασία των οτόκων ορνήθων. Εγώ νομίζω πρέπει να μιλήσουμε και για τα οικονομικά συμφέροντα. Εγώ είμαι Γερμανίδα και εσείς γνωρίζετε. Εμείς ήμασταν χώρα Εξαγωγό αυγών, τώρα έχουμε γίνει εισαγωγό, εισαγωγέ ε, ε, αυγών. Τα, αυγά προέρχονται από κότες που βρίσκονται μέσα σε κλωβούς. Οι καταναλωτές μας πιέζουν ωστόσο, γιατί θέλουν να διατηρηθούν οι τιμές. Μιλήσατε για έναν αριθμό, έναν ορισμένο αριθμό εκμεταλλεύσεων που διαθέτουν κλωβούς. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας αριθμός χωρών μελών που δεν έχουν πράξει το καθήκον τους. Γιατί λέτε ότι από το 1999 τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχουν δοθεί σαφείς εντολές. Εγώ νομίζω ότι βέβαια οι εκκλήσεις δεν αρκούν πλέον. Πρέπει κανείς να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ θα ήθελα πολύ να το πράξετε αυτό Προ το συμφέρον των χωρών εκείνων μελών οι οποίε έπραξαν το καθήκον του, αλλά και βεβαίω και προ το ε, συμφέρον των ίδιων των ορνήθων όσο και των καταναλωτών. Τώρα για το μέλι, το είπατε και εσεί, το θέμα δεν είναι απλό. Η επισήμανση κατά πάσα πιθανότητα ακόμα και αν γίνει δεν θα είναι επαρκή. Νομίζω ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερε επιστημονικέ μελέτε και για την συνύπαρξη και, και με, με γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Λοιπόν θα χρειαστούμε επιστημονικές μελέτες για να μπορούμε να έχουμε σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία. Έχω και μια παράκληση. Το πρόβλημα της διοξίνης στον τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, τι μπορείτε να κάνετε εσείς, έτσι ώστε να ζητήσουμε από όλες τις χώρες μέλη εδώ να θεσπίσουν και να τηρήσουν σαφείς και διαφανείς κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, εδώ μάλλον δεν θα ήμουν σε καμία περίπτωση κατάλληλη να αναλάβω τη θέση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου. Τι θα έκανα, σκεφτόμουν το πρωί αν ήμουν ο ε, Επιτροπός Νταλή και έπρεπε να πάω στο άντρο του Λόντων, το Ευρωκοινοβούλιο που μόλις το 2010, το Σεπτέμβριο συγκεκριμένα, ζήτησε τις υπηρεσίες, από τι υπηρεσίε να, Επιτροπή να, να μας πούνε τι κάνετε για το θέμα αυτό. Η απάντηση δεν ήταν ικανοποιητική. Υπήρχε ψήφισμα από τον Δεκέμβριο του 2010. Το συμπέρασμά μου λοιπόν ήταν ότι θα, αν ήμουν επίτροπος θα τολμούσα να μπω στο άντρο αυτό μόνο στη φωλιά του λύκου, μόνο αν είχα κάτι να πω. Κάτι που δεν είχαμε ξανακούσει τέλο πάντων. Η μόνη κραυγή που έρχεται από τη δική μας Επιτροπή είναι πείτε μας τι συγκεκριμένα θα κάνετε, τι συγκεκριμένη δράση. Ακούμε πολύ ωραία λόγια για επιπαραβάση διαδικασίες. Όμως το να ξεκινούν να κροάσει το 2012 μόλις, τι σημαίνει, ότι έχετε συνολική εικόνα ήδη. Όχι. Εάν ε, αρχίσει κάτι μέχρι το 2012, αν το έχετε πάρει χαμπάρι, θα είμαστε τυχεροί. Και η επιπαραβάση διαδικασία θέλει 1,5 χρόνο για να ακουστεί η πραγματικότητα. Τι λέμε τώρα, το 2014? Τότε θα αποφασίσετε αν θα τιμωρήσετε ένα κάτω μέλος ή τον, ε, ούτε καν όμω τον ε, συγκεκριμένο παραγωγό δεν θα πιάσετε, που δεν έχει εφαρμόσει του κανόνε του οποίου είχε από το 99 για να του εφαρμόσει. Ε, με συγχωρείτε αν δεν έχω εντυπωσιαστεί από το έργο σα και τα λόγια σα, αλλά αυτά περί διαδικασία δεν μα λένε τίποτα. Οι παραγωγοί γελάνε. Το μόνο συμπέρασμα είναι ότι οι παραγωγοί που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει του κανόνε, από όλο αυτό αν δεν μου επιτρέπετε το φιάσκο, τι θα έχουν συμπεράνει. Ότι μπορούμε να κάτσουμε στις καρέκλες μας και να ξαπλώσουμε και να μην ακούμε καν τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μα δώσουν και άλλα τρία-τέσσερα χρόνια για να υλοποιήσουμε στην πράξη τι συμβαίνει. Αυτού τιμωρείτε. Όχι. Αυτού που έχουν εφαρμόσει του κανόνε τιμωρείτε. Αυτού που ήδη έχουν αυξήσει το κόστο τη παραγωγή του από 8 έω 13% σε σχέση με τα συμβατικά αυγά. Η παραγωγή λοιπόν αυτή, αν έπρεπε να του δώσω εγώ κάποια συμβουλή, θα ήταν άστατο την άλλη φορά. Καλύτερα περιμένετε. Κάντε ότι και οι Βέλγοι, που του δώσαν κι άλλο ένα χρόνο. Είναι θέμα λοιπόν αξιοπιστία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να μου πείτε, και εμεί αυτό ζητάμε να ακούσουμε. Το είπαμε με σαφήνεια στο ψηφισμά μα και πάλι αρνείστε να απαντήσετε. Θέλουμε να ακούσουμε τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε με αυτά τα εκατομμύρια αυγά. Από την 1η Ιανουαρίου δεν θα έχουν παραχθεί βάσει των κανόνων. Θα πολλούνται κανονικά. Μήπω θα πολλούνται κανονικά εντό του κράτου παραγωγή. Τι ετικέτα θα έχουν. Τι θα κάνετε με τι εισαγωγέ από τρίτε χώρε. Αυτά τα ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα. Η Επιτροπή μας μπούχτισε, μπούχτισε και βαρέθηκε να ακούει αυτές τις ωραίε δηλώσεις, αλλά να μην βλέπει καμία δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Ντάλη. Θα δούμε αν πραγματικά αξίζεται συγχαρητήριων μετά την εννιαετία που πέρασε και τι αλλαγές είχαμε στην πράξη. Είναι μια από τις λίγες φορές που δοκιμάζεται στα όρια της η κοινοτική νομοθεσία. Και το θέμα είναι αν θα εφαρμόσει την κοινωτική νομοθεσία ή μπορεί κανείς ατιμόρυτα να την παραβιάζει, να την αγνοεί. Και το θέμα των οτόκων ορνήθων είναι σήμερα αντικείμενο συζήτηση. Αλλά θα έχουμε και άλλα προβλήματα μέσα σε ένα χρόνο. Την οδηγία για τους χείρους που θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Πρώτου 2013. Τι θα συμβεί εκεί. Θα έχουμε ε, καλύτερη ζωή πραγματικά από την 1η Πρώτου του 2013 ε, για τα γουρνόπουλα και τους ε, χείρους ή θα συνεχίσουν οι άθλιες ηθίκες διαβίωσης στη χειροτροφία. Είμαστε Επιτροπή Γεωργίας και θα πρέπει να είμαστε και διορατικοί. Μην ξεχνούμε τους χείρους. Επειδή αποσπά την προσοχή μας αυτή τη στιγμή από τις κότες και τα αυγά. Υπάρχουν προτάσεις ε, για μια νέα στρατηγική για την περίοδο 2011-2015. Αλλά σχεδόν έχει εκπνεύσει το 2011 και στρατηγική δεν έχουμε δει ακόμη. Ευχαριστώ ο κύριος Πόλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είμαι ακανακτισμένη. Μας είπατε τα ίδια πράγματα που μας είχατε πει προ λίγων μηνών επαναλαμβάνεται τα ίδια πράγματα για τα αυγά και νομίζω ότι δεν έχετε περιλάβει απολύτως κανένα στοιχείο. Γνωρίζουμε ότι από 1η Πρώτου 2012 θα αρχίσει η απαγόρευση. επίση επίσης ότι από 1η Πρώτου 2012 θα υπάρχουν εκατομμύρια παράνομα αυγά στην αγορά. Και λέω παράνομα διότι δεν θα ανταποκρίνεται η παραγωγή τους στην νομοθεσία μας. Ξέρουμε ότι θα υποβάλλεται και θα ξεκινήσετε διαδικασίες παραβιάσεως. Αν είμαι επιχειρηματίας όμως, τι με νοιάζει, αφού η εθνική μου κυβέρνηση θα κληθεί να πληρώσει. Θα ήθελα από αυτού να μου απαντήσετε. Εν τέλει πόσα εκατομμύρια αυγά, για πόσα εκατομμύρια αυγά μιλούμε. Από 1η πρώτου 2012 θα βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας εικόνες καταστροφής εκατομμυρίων αυγών. Πώς θα τα δικαιολογήσετε αυτά τα πράγματα. Εγώ αναμένω μέγα σκάνδαλο. Πώς θα καταστήσουμε πιστευτά στους ε, πολίτες τα πράγματα αυτά ότι καταβάλαμε προσπάθεια τους τελευταίους μήνες να επιτύχουμε κάποιες λογικές λύσεις. Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν μας παίρνετε στα σοβαρά και ούτε μπορώ να αντιληφθώ πώς θα μας πάρουν οι πολίτες στα σοβαρά εάν συνεχίσουμε να δρούμε με τέτοια αμέλεια. Και για το μέλι τώρα, από Σεπτεμβρίου 2012, λέει ο Μιλήτρια, υπάρχει μία απόφαση και λέει ότι δεν λειτουργεί η συνύπαρξη αυτή γάματα φόμικρων και μελιού. Θα συνεχίσετε να, να επιτρέπετε την, τις ε, εσοδίες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη ή θα προστατεύσετε επιτέλους το μέλι. Και πώς θα εξασφαλίσετε στους καταναλωτές το δικαίωμά τους να καταναλώνουν μέλι χωρίς προσθήκες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ελπίζω να λάβω απαντήσεις. Ευχαριστώ, Μολυκέ. Ο Τζιμ Νίκολσον και μετά ο Πετραγιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήμουν ε, καλός με τον Επίτροπο, που θα ήταν αλλαγή μετά από τόσα που το έχουμε πετάξει. Τέλος πάντων, θα πρέπει όμως κάπως να προχωρήσουμε. Διότι όλοι οι Βρετανοί μέλη αυτής της Επιτροπής από την ε, περασμένη εβδομάδα έχουν λάβει τουλάχιστον 6.000 mail. Τέλος πάντων οι βοηθοί μας, όχι εμείς οι ίδιοι μόνο. Ε, το ίδιο που έχουμε ακούσει τόσες φορές. Υπάρχει τεράστια ανησυχία, Επίτροπε. Δεν θέλω να επαναλάβω σε επανεπροελίσσαντες. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι θα υπάρξουν περίπου 80 εκατομμύρια αυγά την 1η Ιανουαρίου που δεν θα έχουν παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα είναι παράνομα. Τι θα κάνετε, τι θα συμβεί με τα αυγά αυτά, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πολύ γεωργοί και εκτροφείς έχουν κάνει σοβαρότατες επενδύσεις προκειμένου να, φτάσουν τις, να αναβαθμίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να φτάσουν στα πρότυπα που τους απαιτούμε να σέβονται. Έχουν πολύ επιπλέον κόστος για να παράγουν τα αυγά τους. Τι θα κάνουμε, τι θα πει. Τι θα πει ότι θα στείλετε τους ανθρώπους σας στις διάφορες χώρες. Ποιοι είναι αυτοί που θα εντοπίσουν τα αυγά. είναι συγκεκριμένα άτομα, μήπως πρέπει να μάθουμε και την ταυτότητά τους. Και όταν λέτε ότι θα στοχεύσουμε συγκεκριμένα κράτη, τι θα πει με τη, ότι θα κάνετε με τη διαδικασία επί παραβάση. Μέχρι το 2014 φαίνεται ότι θα κρατήσει όλη η διαδικασία. Πώς θα πάψουν αυτοί οι άνθρωποι να παράγουν και τι θα γίνει με αυτά που εξάγονται, εξάγονται εκτό συνόρων εφόσον έχουν παραχθεί παράνομα. Και τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη που για να υπερασπιστούν τους παραγωγούς τους θα αναλάβουν δική τους δράση μόνοι τους, θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές αυγών. Ε? Κύριε Νίκολσον, σας ευχαριστούμε. Όλοι φαίνεται ότι έχετε εξαντλήσει την εμπνευσή σας κατά το Επιτρόπου Νταλή σήμερα. κατευθείτε για την επόμενη με τον κύριο Σιόλο, ο Πέτερ Γιάρτορα. Ε, ε- Και μετά, κυρία Έραν Διακυβεύεται η αξιοπιστία μας, διότι πρόκειται πολύ απλά. Οι νόμοι που φτιάχνουμε εδώ εφαρμόζονται. Για σκεφτείτε το αντίθετο. Διότι καθόμαστε εδώ και μαλώνουμε για κανονισμούς, για οδηγίες, νομοθετούμε και μετά δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ο κανονισμός για τις συστοιχίες κοβών ορνήθων είναι κακό παράδειγμα. Είχαμε 12 χρόνια για την για να περάσουμε στην εφαρμογή. Δεν πρόκειται για κανένα αναπάντεχο φαινόμενο και προφανώς ουδής ασχολήθηκε. Κανένα δεν ενδιαφέρει η νομοθεσία αυτή. Εμείς και επομένως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεχθήκαμε αυτό. Ξεκινήσαμε ένα monitoring πριν από μία διετία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε πει ότι ναι, θεωρούμε ότι όλες οι χώρες θα αρχίσουν ταυτόχρονα την εφαρμογή της απαγορεύσεως. Σε ορισμένες περιφέρειες φαίνεται ότι αυτό είναι αδύνατον. Γιατί δεν έγινε σωστά το monitoring και έρχεται τώρα το ερώτημα τι θα κάνουμε την πρώτη μέρα εφαρμογής ε, η συνάδελφός μου Ντελάνζ είπε για τις χώρες μέλη ότι θα δράσουν αυτές. Ίσως είναι πολύ αισιόδοξο. Εγώ βρίσκω ότι αυτά είναι πολύ λίγα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι θα κάνουμε την 1η Ιανουαρίου του 2012 όταν θα αναγκάσουμε εν τέλει τους καταναλωτές μας να καταναλώνουν αυγά τα οποία έχουν παραχθεί παρανόμως. Περί αυτού πρόκειται. Δεύτερο, για το, για το μέλι. Εκεί σωστά είπατε ότι τα προβλήματα αποτιθείται είναι κυρίως πρακτικού χαρακτήρα. Η ερώτησή μου είναι μήπως κάναμε λάθος. Που λέμε, μου κάνει ε, τη διάκριση η ε, απόφαση ανάμεσα σε φυτονομικά προϊόντα και σε τρόφιμα. Και τι θα κάνουμε με τις ανεξάρτητες αποφάσεις των χωρών μελών. Οι μέλισσες όμως δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι μέλισσες θα περάσουν από τα σύνορα και θα πάνε από τη Γερμανία στην Τσεχία. Τέλος, για τις οριακές τιμές. Πρέπει να εξετάσουμε οριακές τιμές, ναι ή όχι. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρας Γκαρσία και μετά ο κύριος Ντές, κατόπιν η κυρια ρας Μαγκίνας. κυριος δες Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε να μας εξιστορίσετε αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Φαίνεται ότι εμεί δεν έχουμε τίποτα να καταφέρουμε. Οι Ισπανοί παραγωγοί είχαν ζητήσει παράταση μέχρι το 2014 γιατί δεν προλάβαιναν να εφαρμόσουν τι διατάξει για τέτοιου είδου κλοβού. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει τέτοια παράταση, αλλά θα ευνοηθούν εδώ όχι τελικά οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ, αλλά χώρε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Βραζιλία, που θα εξαγάγουν ε, άπειρα αυγά προς εμάς, από αυγά από κότες που βρίσκονται σε, διαβιούν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τις στοιχείες κλωβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, πώς θα αποφύγουμε είτε τα εισαγόμενα αυγά να παράγονται σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι στην Ευρώπη, οπότε έτσι εξηγούνται τα αυστηρά μετρελέχου που επιβάλλεται στα κρατημέλη, ή πώς θα αποφύγετε ε, τον τάμπιξ τιμή των αυγών ε, ή ε, αν δεν έχουμε εισαγόμενα αυγά να εκτιναχθούν οι τιμές των τόπιων αυγών στα ύψη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε άριστη κατάσταση των εισαγόμενων αυγών. Γιατί πώς θα εξηγήσουμε στους ε, Ευρωπαίους πολίτες που όλο και υφίστανται μέτρα λιτότητα ε, ότι εφαρμόζουμε τέτοιου είδου μέτρα. Επίση, υπάρχει υποχρέωση άδεια ανεξάρτητα από την ε, προέλευση του περιλαμβανόμενου στο προϊόν γενετικώ τροποποιημένου στοιχείου. Τι ε, μέσα θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί θα κατακλειστείτε από τέτοιε αιτήσει. Στην Ισπανία το 80% της επικράτειας είναι ανοιχτό για γενετικό τροπημένους οργανισμούς, οπότε το μέλι που παράγεται στην Ισπανία θα για το μέλι που, παράγεται στην Ισπανία θα ζητηθεί μαζικά τέτοιου είδους ε, άδεια τι μέτρα θα θες, θα χρησιμοποιήσετε και θα πώς μπορείτε να διευκολύνετε τους γεωργούς. Τίποτα δεν είπατε για τα συμπεράσματα της α, ε, σύσκεψης που είχαν εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στην ε, Ειδική Επιτροπή για την Τροφιμική Αλυσίδα, θα μέσα του Σεπτεμβρίου. Ποια είναι τα συμπεράσματα αυτής της σύσκεψης των εμπειρογνωμόνων. Έχετε κάποια στοιχεία να μας αναφέρετε. Ο Άλμπερτ Ντες και μετά κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, πολλοί από τους συναδέλφους μου διαμαρτύρονται ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται εδώ δεν είναι αρκετά γρήγορες. Εφτά χρόνια είμαι ευρωβουλευτής, τα τελευταία χρόνια μίλησα αρκετές φορές μαζί σας και παρόλη την κριτική που ακούστηκε σήμερα θεωρώ ότι μπορώ να σας επενέσω, διότι είστε ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει δράση όταν αυτό είναι απαραίτητο. Υποθέτω ότι και τώρα στη δύσκολη αυτή υπόθεση των οτόκων ορνήθων αλλά και του μελιού θα βρείτε τις σωστές απαντήσεις. Και ελπίζω ότι και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε για να εξεύρουμε τις ορθές λύσεις. Λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρηθούν. Όπως είπαν άλλοι συναδελφοί μου, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν υπέρεπαρκής. Έπρεπε να είχαν προχωρήσει περισσότερα τα πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Κάποια συγκεκριμένα ερώτηματα. Για τα αυγά που θα παράγονται σε συμβατικό και θα μένουν εκτός πωλήσεων από 1η Ιανουαρίου 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περιορίσει το εμπόριο των αυγών αυτών και πώ θα το κάνετε. Τρίτο. στοχεύοντα κάτι μέλη, θα στοχεύετε αυτούς που συμμορφώθηκαν ή τους ασυμμόρφωτους. Διότι άμα ξεκινήσετε με τους άτακτους και τους ε, ανυπότακτους θα μας πάρει καμιά δεκαετία. Μήπως να κάνετε το ανάποδο λοιπόν. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, αλλά νομίζω για τους παραγωγούς που έχουν επενδύσει για, τα, για τις εμπλουτισμένες κλωβούς, εκείνοι θα στραφούν εναντίον μας, εάν επιτραπεί στους υπόλοιπους να εμπορεύονται Κατάλαβα Τι, τι, να πω για του Ισπανού συνάδελφου που λένε ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Απαντήστε παρακαλώ στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Λεμπρεν. Η κυρία Λεμπρεν, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να ενώσω εγώ τη φωνή μου στη χοροδία αυτή της αγανάκτηση. Ήταν αρκετά βολονταριστικά τα σχόλια του Επιτρόπου, αλλά θα ήθελα να προσθέσω στον ναι μεν το ένα αλλά, γιατί υπάρχει το αλλά. Ε, είχαμε ένα αντίκτυπο για την ενιαία αγορά. Πολύ σημαντικό αυτό το μέσο και σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε και την παρούσα κρίση. Σίγουρα η εναρμόνιση των κανόνων ίσω ε, δώσει όθηση για την ανάπτυξη. Εν αυτή την ποιο θα είναι το μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πλήττοντα του παραγωγού που συμμορφώνονται με την ενιαία αγορά σε σχέση με αυτού που δεν τη σέβονται. Μία από τι ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν να ε, δράσει πραγματικά ως θεματοφύλακας της ηθίκης. Καταλάβαμε ότι θα δείξει πυγμή ε, η Επιτροπή απέναντι στα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται. Αρκούν όμως ε, απλές απαντήσεις. Περιμένουμε κι εμείς, όπως είπαν οι συνάδελφοι, σαφή μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, η πατρίδα μου, η δική, η δική μου πατρίδα έχει συμμορφωθεί με την κοινοτική νομοθεσία και η, παραγωγή, εθνική παραγωγή μειώθηκε κατά 8%. Ενώ άλλε χώρες που δεν συμμορφώθηκαν αύξησε την παραγωγή τους κατά 16%. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη και τυπικά και ουσιαστικά να αποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί πραγματικά να ασκήσει το ρόλο της ως εκτελεστικής εξουσίας. Είτε θεσπίζοντας σαφείς στους συγκεκριμένους και κατηγορηματικούς κανόνες, είτε βοηθώντας τους παραγωγούς ή τις χώρες που ήδη συμμορφώθηκαν με τους κανόνες. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να προσθέσω κι εγώ ότι εμείς ε, στις εκλογικές μας περιφέρειες, στις πατρίδες μας ε, έχουμε προβληματιστεί γιατί μας έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και πλησιάζουμε σε μια έκριθμη κατάσταση που μπορεί να ξεσπάσει και σε σκάνδαλο αν δεν έχουμε άμεσα κάποια μέτρα πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε δέκα ακόμη ομιλητέ. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο αγόρευση ο καθένα. Ο κύριο Χάουσλινγκ. Κύριε Επίτροπε, ε, να μην ξαναμιλήσω κι εγώ για τα αυγά, γιατί αρκετά μιλήσαν άλλοι. Μία ερώτηση μόνο. Πεςτε μας καθαρά ποιες είναι οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρώσεις τους. Και είναι αληθές ότι ορισμένες χώρες δεν έχουν δώσει απολύτως καμία πληροφορία. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να το ξέρουμε. Τώρα για το μέλι. Σωστά περιγράψατε την κατάσταση. Στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει πώς θα μπορέσει να εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου. Και η ερώτηση που έχω είναι, μιλήσατε πολύ για ελέγχους του μελιού αλλά αυτό στην ουσία σημαίνει ανάγκη μεταρρύθμισης των ε, κανόνων για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε απαγόρευση πτήσεων στις μέλισσες, αλλιώς το μέλι που θα φτάνει στην αγορά είναι παράνομο. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε εισαγωγή παντός είδους μελιού αυτή η δίθεν μηδενική ανοχή σας δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί. Διότι μηδενική ανοχή σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει απολύτως καμία, κανένα ίχνος μάλλον γύρισα από ε, τροποποιημένους οργανισμούς στο μέλι. Ο κύριος Αγνιό και μετά Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Κύριε Πρόεδρε, αρχίστε να με χρωματείτε από τη στιγμή που θα αρχίσει να με κοιτάζει ο Επίτροπος. Περίμενα κάτι χρήσιμο από εσά σήμερα, κύριε Επίτροπε. Ήταν σκληρά τα μέτρα, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Το μόνο που κάνατε είναι ότι θα μα υποσχεθήκατε ότι θα έχουμε φορτηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βγάζει τα αυγά εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα σπάει. Δεν πρόκειται να το κάνετε δεν νομίζω ότι τα μέτρα αυτά θα είναι αποτελεσματικά. Θα πάτε σε καμία μονάδα, ε, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει συμμόρφωση, υμόρφωση υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχει συμμόρφωση. Και το θέμα των αδειών είναι προβληματικό, ακόμη και όταν εφαρμόζονται για τις στοιχείες κλωβών. Μπορείτε να με κατηγορήσετε ε, ότι είμαι φιλοβεωρετανός, αλλά φυσικά αυτό που θέλω είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της κυβέρνησης και να πιεστούν οι εισαγωγείς να ασκήσουν τον δέοντα έλεγχο στην εισαγωγή αυγών. Έχουμε 25-30 διαφορετικές αλυσίδες ε, ελληνικού εμπορίου. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ε, εντοπισμός προέλευσης των αυγών και να κατονομάζονται οι λιανέμποροι που παραβιάζουν τις ε, διατάξεις. Νομίζω το οφείλουμε αυτούς τους κατανοτές της Μεγάλης Βρετανίας. Κυρία Ρέιμερς ούτω ή άλλω μιλάω πολύ γρήγορα, θα προσπαθήσω να μιλήσω τόσο γρήγορα, για τι ε, συστοιχίε κοβών ορνήθων. Μιλούμε διαρκώ για παράνομα αυγά, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται, πρέπει να μιλάμε για παράνομε κότε. Εάν ο κλοβός είναι παράνομο, τότε είναι παράνομη και η κότα που βρίσκεται μέσα πριν να φτάσει να γίνει το παράνομο αυγό. Πώ θα απελευθερώσουμε τι παράνομε κότε από τα παράνομα κλουβιά, Αυτό είναι το ερώτημα. Και αυτό σημαίνει είδατε ότι έχετε μεγάλη υποστήριξη από εμάς να προχωρήσετε ενεργά, δραστήρια απέναντι στις χώρες που δεν τηρούν τις υποχρώσεις τους. Διότι υπήρξε επαρκής χρόνος, μεγάλη μεταβατική περίοδος, ασυνήθιστα μεγάλη. Και μάλιστα δόθηκαν και, και χρήματα για υποστήριξη για τις τροποποίησεις. Δόθηκε λοιπόν υποστήριξη στις επιχειρήσεις οι οποίες άλλαξαν τις μεθόδους παραγωγής. Άρα λοιπόν δεν θα δώσουμε στο μέλλον χρήματα για να υποστηρίξουμε άλλες επιχειρήσεις. Έχετε το θάρρος να σφραγίσετε, να κλείσετε τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες δεν τήρησαν τις υποχρώσεις τους. Και για το μέλλον, Δεν είναι πλέον ούτε καν 12 και 5, είναι 12 και 20 σε ό,τι αφορά την ανάγκη ρύθμισης, νομοθετικής ρύθμισης για τη λεγόμενη συνύπαρξη. Μιλούμε μόνο στην Ευρώπη για μηδενική ανοχή. Ενώ ταυτόχρονα δεχόμαστε τα τρόφιμα που εισάγονται σε μεγάλο βαθμό να έχουν προκύψει από συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και ε, της παραγωγής τους. Πρέπει να δούμε ότι, πρέπει να δούμε ότι εκεί υπάρχει ανάγκη μάλλον να γίνει κάποια ε, πρόοδος. Σμιτ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν άλλοι συνάδελφοι. Θα συμφωνήσω με τον Τζιμ Νίκολσον και θα είμαι και εγώ συμπαθητικός απέναντι στον Επίτροπο. Αλλά μην παρανοήσετε τα λόγια μας γιατί έχουμε μεγάλη απογοήτευση από την έλλειψη δράσης που βλέπουμε. Όλες και όλοι μας εδώ έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε τις ε, κοινοτικές ρυθμίσεις απέναντι στους γεωργούς μας και στους πολίτες μας. Και έχουμε και τις δυσκολίες που γνωρίζετε και με την ηλεκτρονική επισήμανση των προβάτων στη Σκοτία κλπ. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες αυτούς. Τώρα, για το μέλι. Είναι ηθικός ο κίνδυνος και για τις ε, όρνηθες. Εάν δεν επιτύχουμε να εφαρμόσουμε τις ρυθμίσεις αυτές, θα πάψει να ενδιαφέρεται ο κόσμος, δεν θα έχει καμία εμπιστοσύνη απολύτως. Θα έχουμε βέβαια κάποιες διαδικασίες παραβίασης στο μέλλον, αλλά αυτά τα πράγματα είναι και πολύ καθυστερημένα και πολύ λίγα. Χρειαζόμαστε να σταματήσουν οι υποστηρίξεις, χρηματοδοτικές υποστηρίξεις στους παραγωγούς αυτούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να παράγουν με τρόπο παράνομο. Σας ζητούμε λοιπόν να αναλάβετε αυστηρότερη δράση απέναντι σε χώρες μέλη. Εγώ νομίζω ότι είναι ανεύθυνο να καταστραφούν τέτοιες ε, μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Δεν λέω να τα σπάσετε τα αυγά, αλλά θα επανέλθω σε ένα ερώτημα. Αφού το προϊόν αυτό θα είναι παράνομο μετά από την πρώτη του έτους, τότε οι χώρες μέλη οι οποίες θα κλείσουν τα σύνορά τους στις εισαγωγές τέτοιων παράνομων τροφίμων είναι, συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και για το μέλη τώρα οι μελέτες που έχετε ζητήσει μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε αναδρομικά να, γίνουν, να, να δοθούν οι άδειε εισαγωγή. Και τέλος, τι μήνυμα είναι αυτό που δίνεται στους παραγωγούς γενετικά τροποποιημένων ε, τροφίμων και ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποζημίωση των παραγωγών. Ευχαριστούμε κύριο κύριος και μετά κύριο κύριος Μποβέ. Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα και ευχαριστούμε που μας είπατε αυτό που έπρεπε να μας πείτε. Δηλαδή ότι από 1η Ιανουαρίου του 2012 αρχίζει να ισχύει ο νέος κανονισμός και ότι όποιος δεν προσαρμοστεί, δεν συμμορφωθεί, θα τιμωρηθεί. Αυτό έπρεπε να μας πείτε και μας το είπατε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κι εγώ κάτι. Προαναγγείλατε ότι με μεγάλη αποφασιστικότητα και δυναμισμό θα πράξετε το δέον ότι θα ακολουθήσετε τους νόμους και κανόνες. Όμως, κάποιες ευκαιρίες πρέπει και αυτές να τις ε, σκεφτούμε. Όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες, μπορεί να μην το έκαναν μόνο επειδή δεν τους άρεσαν οι κανόνες, αλλά δεν μπόρεσαν να συμμορφωθούν. Κάποιοι λοιπόν δεν ακολούθησαν τους κανόνες όχι για να ξοδέψουν τα ίδια χρήματα σε άλλες επενδύσεις, γιατί οι δυσκολίες της αγοράς ή οι τιμές των προϊόντων ε, βρίσκονταν σε μείωση. Η Ευρώπη λοιπόν τι θα κάνει, θα επιβάλλει περισσότερες κυρώσεις στους παραγωγούς αφού όποιος δεν καταφέρει να συμμορφωθεί με τους κανόνες, ε, μάλλον αν θέλουμε να πετύχουμε τέλεια αποτελέσματα θα πρέπει να πάψει την παραγωγή του ποιος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες. Τι θα γίνει όμως, ε, θα ξεχάσουμε τους παραγωγούς αυτούς που έχουν προβλήματα οι κότε θα φύγουν, θα πάνε στις χώρες εκτό Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι συνθήκε θα επιδεινωθούν πάρα πολύ σε σχέση με τις τωρινέ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τέλος πάντων αυτές που αφορά ο νέος κανονισμός. Τώρα προκύπτει και ένα άλλο στοιχείο. Η τελο παντων αυτες που αφορα ο νεο κανονισμο τωρα προκυπτει και ενα χτυπά την αγορά, την κατανάλωση και την ίδια την παραγωγή. Θέλουμε με σιδερένια γροθιά να αναλάβουμε δράση επίτροπε Πρέπει να γίνει και αυτό, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σκόπιμο. Περαιτέρω μέτρα που να επιτρέπουν περαιτέρω κανόνες που να επιτρέπουν την εμπορία των αυγών αυτών ή ε, έστω στο εσωτερικό της χώρας παραγωγής τους όταν πρόκειται για εκμεταλλεύσεις ε, που δεν έχουν καταφέρει να συμμορφωθούν με τους κανόνες, αυτό επίτροπο πρέπει να το προβλέψουμε. Εντάξει, αυστηρότητα για την υλοποίηση του κανονισμού, αλλά δείτε τι έγινε τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια. Χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα. Η συνάδελφος που πήρε το λόγο προηγουμένως είπε ότι πολλοί πόροι τέθηκαν στην υπηρεσία της στήριξης με οικονομικές επενδύσεις στην αλλαγή των κλοβών συγκεκριμένα. Όμω, Επίτροπε, χρειάζονται και άλλα κονδύλια εδώ και άλλοι πόροι. Κάποιοι δεν κατάφεραν να το κάνουν ω τώρα, να του βοηθήσουμε. Ολοκληρώνω, Επίτροπε, απευθύνοντας έκκληση πέραν των λόγων των νομοθετικών να σκεφτείτε και τους ε, λόγους της σκοπιμότητας. Σήμερα κυρώσεις επιπλέον θα πλήξουν και θα γονατίσουν τους παραγωγούς μας. Αυτοί που θα ωφεληθούν είναι παραγωγή εκτός Ευρώπης. Αυτοί με όρους και πρότυπα πολύ λιγότερο ασφαλή θα έρθουν για να ανταγωνιστούν τις δικές μας τις κότες. Ο κύριος Μποβέ και μετά ο κύριος Λάιον. Κύριε Επίτροπε, Δεν συνηθίζω να σας συγχαίρω, αλλά σήμερα θα το κάνω. Γιατί πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δράσει υπέρ της ευημερίας των ζώων. Γιατί πολύ συχνά μιλούμε για αυγά και για προϊόντα εκμετάλλευσης, αλλά αγνοούμε τα ζώα. Και το μέτρο αυτό ψηφίστηκε προκειμένου να βελτιωθεί ε, η κατάσταση στην κτηνοτροφία υπέρ της ευημερίας των ζώων και νομίζω ότι ε, το δικό τους συμφέρον προσπίζουμε με τη διάταξη αυτή. Προσοχή όμως, να έχουμε σαφή εναρμόνιση για τα εισαγόμενα προϊόντα. Γιατί θα ήταν πραγματικά παράλογο και ανώμαλο να έχουμε μια πρακτική συγκεκριμένη δεδομένη εντό Ευρώπης και τα εισαγόμενα προϊόντα να μην υπάγονται σε αυτούς αυστηρούς κανόνε. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι λοιπόν πιο απαιτητική εναρμόνιση στι αγορέ και όχι μόνο εσωτερική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο σχόλιο για του γενετικώ τροποποιημένους οργανισμού. Τρει απλούστατε ερωτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια σκέψη και μια ιδέα για την ρήπανση των, της γύρης και των, του μελιού στην Ευρώπη ή πώς θα προβεί σε μια τέτοια αξιολόγηση της α, αυτή. Ε, ρήπανσης αυτής. Γιατί αναφέρθηκε το καλαμπόκι 810. Αλλά Έχουμε και ρήπαση από γύρι ελοκράμβης, βαμβακιού και άλλων φυτών και ίσως εκεί δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί αυτές οι φυτίες, ε, καλλιέργειες δεν επιτρέπονται στην Ευρώπη. Αλλά μπορούν να προέλθουν από άλλη χώρα. Από τη στιγμή που εμάς τις απαγορεύουμε θα πρέπει να απαγορεύουμε και την εισαγωγή. Και ένα πρόβλημα που ανακύπτει με την νομοθεσία θα πρέπει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβει μια πιο περίφραστη θέση. Τρίτον, δεύτερον, συγγνώμη, τι αντισταθμιστικά μέτρα θα θεσπίσετε σε περίπτωση απαγόρευση του αποχαρακτηρισμού της γύρης και του μελιού για τους μελισσοκόμους, γιατί αυτοί θα πληγούν από την μόλυση που δεν την επιδίωξαν. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να ενημερώσει τους καταναλωτές για τα εισαγόμενα μέλη από την Αργεντινή, για παράδειγμα πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν σφραγίδε στο μέλι αυτό, μέλι με γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού, για να έχουν δικαίωμα επιλογή οι καταναλωτέ να γνωρίζουν τεκμηριωμένα τι μέλι αγοράζουν, αν περιλαμβάνει γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού ή όχι. Ο κύριο Λάιον και μετά Λάντερφελτ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μη τι άλλο μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες προς τον Επίτροπο Ντάλι που τουλάχιστον ήρθε ε, και αντιμετώπισε ε, μόνος του την ε, κατακραυγή και δεν στείλετε κανένα υπάλληλο για να υπερασπίσει τα απαράδεκτα μπροστά μας. Αν μη τι άλλο γι' αυτό, σας αξίζουν συγχαρητήρια. Υπάρχουν πολλά θέματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Εμείς, ως ευρωβουλευτές που ε, σας επισημάναμε όλα αυτά τα πράγματα, με τι μούτρα θα γυρίσουμε στους καταναλωτές και τι θα τους πούμε. Τι θα τους πούμε ότι θα συμβεί από την 1η Πρώτη του 2012. Τι θα πούμε στον ε, Γεωργό που έχει επενδύσει 10 εκατομμύρια ε, στερλίνες λίρες για ε, ε, να καταργήσει τους κλοβούς και να αφήνει τις ε, κότες του να, να βόσκουν ελεύθερα. Πώς θα το δικαιολογήσουμε όλα αυτά. Γιατί θα έχουμε εισαγόμενα αυγά που δεν θα ξέρουμε καν ποιος θα παράγει αυτά τα παράνομα αυγά. Νομίζω ότι έτσι απαξιώνεται ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο, οι ευρωπαϊκές διατάξεις, η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ποιος παραγωγός που δεν συμμορφώθηκε θα σπεύσει να συμμορφωθεί μια και δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης. Δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Ξανασκεφτείτε το θέμα αυτό και υποβάλλετε πραγματικά ένα σχέδιο με πυγμή που θα υποχρεώσει τους παραγωγούς να συμμορφωθούν και οι καταναλωτές από την πρώτη πρώτη να ξέρουν ότι τα αυγά που καταναλώνουν ε, έχουν παραχθεί σε, κλωβού, σε κλωβούς που σέβονται την ευημερία των ζώων. Μόνο με τέτοια μέτρα ε, θα ήταν σωστή η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος ε, Νταντά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχω μια ερώτηση για το μέλι. Η εφαρμογή της ε, σχετικής δικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου μπορεί να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση ό,τι αφορά τη συσκευασία μελιού, που καταναλώνεται όμως από τον Ευρωπαίο καταναλώτη και μπορεί ίσως να οδηγήσει και σε παραπίση νόθευση μελιού. Γιατί υπάρχει μια πλούσια τεχνική, αφαιρείται η γύρη από, τη μέλη, από το μέλι, ενώ ε, η γύρη αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανιχνευσιμότητα του μέλιου. Οπότε θα μπορεί οποιοδήποτε ε, παραγωγός να αφαιρέσει τη γύρια από το μέλι που θα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως μέλι κάτι που θα οδηγήσει σε απώλεια κεφαλαίου παραγωγής και θα οδηγήσει σε, απάτη, σε εξαπάτηση, ε, σε παραπλάνηση μάλλον, συγγνώμη, τον καταναλωτή δεν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία του μελιού ώστε να λάβει υπόψη την ε, γνωμοδότηση της 23ης ε, Ιουνίου του 2004 των εμπειρογνωμόνων που λέει ότι ε, το μέλι δεν εμπίπτει στον κανονισμό 1829 του 2003. Αυτά και λυπούμε δεν θα ακούσω την απάντηση γιατί πρέπει να φύγω σε άλλη συνεδρίαση. Ο κύριος Μπλάτενφελτ. Ευχαριστώ πρόεδρε η περισσότερη παραγωγή αυγών στην Ουγγαρία χρησιμοποιούν ήδη μεγαλύτερους, μεγαλύτερους κλεβούς. Αναρωτιούνται λοιπόν, θα ακολουθήσει αυστηρά τους κανόνες της η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ ακούσαμε κάποιοι να συνηγορούν υπέρ της μεταφοράς των παλαιών κλεβών στην Ουκρανία, όπου η παραγωγή θα συνεχιστεί με το παλιό ευρωπαϊκό σύστημα. Τα αυγά μετά αυτά στην Ευρώπη θα εισάγονται. Πρέπει λοιπόν να αντιλήσουμε εδώ κάποια διδάγματα. Και ένα από τα βασικότερα είναι ότι ο λόγος για τον οποίο τα οι κλοβοί παλαιού τύπου χρησιμοποιούνται ακόμη για να παραχθούν αυγά είναι γιατί βγάζει κανείς κέρδος από όλο αυτό. Όταν πηγαίνει κανείς σε ένα μαγαζί για να αγοράσει αυγά βλέπει ότι τα συμβατικά παραγμένα αυγά κοστίζουν 15 με 30% λιγότερο. Μην ξεχνάμε ότι σε κάποιε περιοχέ τη Ευρώπη κάποιοι δαπανούν το 15-20% του εισοδήματό του για να αγοράσουν τρόφιμα. Λοιπόν, δεν μπορούν να είναι θύματα αυτή τη διάκριση μεταξύ αυγών που έχουν παραχθεί χωρί πρόβλημα και άλλα που υπόκειται σε αυστηρότερου κανόνε. Εδώ μιλάμε για μια παραποίηση και αν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα ισχύει με τα νέα αυγά, κάποιοι νομίζουν ότι αυτό έχει να κάνει με τη χρήση καυσίμων και την κατανάλωση καυσίμων. Όλα είναι σχετικά. Καλή ήταν η ταχεία λήψη απόφασης, αλλά το θέμα είναι λάβατε υπόψη και τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, διότι οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης των γενετικών τροποποιημένων οργανισμών μας απασχόλησαν ιδιαίτερως και βρήκαμε επιχειρήματα για να περιοριστεί η χρήση τους. Όμως τα λάβατε υπόψη. Μάλιστα. Η κυρία Λούλινγκ για λίγα δευτερόλεπτα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, επειδή ευρωπαϊκούς νόμους σχεδιάζουμε, καλό να θυμόμαστε λίγο ότι κάποιοι από εμά που βιαζόμαστε να μιλήσουμε, κάποιες φορές πιο πολύ ανησυχούμε για τη ζωική υγεία από ότι για την ανθρώπινη. Ναι, ναι, καλά ακούτε. οι άνθρωποι θα ζήσουν τι αρνητικέ επιπτώσεις από την υγεία των ζώων. Καλά, μην ξεχνάμε αυτά για την απασχόληση, την ενεργεία και το καθεξής. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση που αφορά τους μελισσοκόμους. Πιστεύω ότι μερικοί μελισσοκόμοι βιάστηκαν να χαρούν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ιδίω όσοι είναι Εμπαθή κατά των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Τώρα οι βαβαροί μελισσοκόμοι εξυπηρέτησαν τους ε, συναδέλφους τους, θα φανεί. Και θέλουμε να μάθουμε τι θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει την εξακολούθηση της μελουσιουργικής δραστηριότητας στις περιοχές παραγωγής γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει με τις ζώνες αυτές που δεν είναι πολλές, αλλά ποιος θα πουλήσει, ποιο θα πληρώσει μάλλον τις ε, αναλύσεις που πρέπει να γίνουν και τις έρευνες, ποιος θα αποζημιώσει τους ε, μελισσοκόμους για την απώλεια και τη μείωση της τιμής των προϊόντων του, ο κύριο Άσβορτ. Και μετά ο Επίτροπος, ο Επίτροπος Νταλή. Τζο. Ε, επίτροπε, θα κλείσω στο ίδιο ύφος με τον κύριο Νίκολσον, αλλά θα σας προσφέρω τη στήριξή μου. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν το 1999 να επιβάλλουν ε, την ισχύ μεταβατικής περίοδου απαιτώντα από τον βιομηχανικό αυτό το κλάδο να περάσει στους εμπλουτισμένους, στις εμπλουτισμένες Τα κράτη-μέλη εδώ και 12 χρόνια δεν έχουν σεβαστεί τις υποχρεώσεις τους ώστε να πιστούν οι δικοί τους οι παραγωγοί, τέλος πάντων να αναγκαστούν να κάνουν την απαραίτητη μετάβαση. Τώρα ο επιτροπο βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, πράγματι. Και γι' αυτό ε, έχω συμπάθεια. Όπως είχα και για τον ε, Επίτροπο πριν από εσά, Τι θα γίνει με τα αυγά από 1η Ιανουαρίου 2012. Στη δική μου τη χώρα τι θα γίνει με τους παραγωγούς που έχουν επομιστεί το σοβαρό αυτό και έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Εσείς είπατε ότι θα ασκήσετε διαδικασία, θα ασκήσετε προσφυγή κατά των, ε, κατά που δεν συμμορφώνονται. Επίτροπε, τι θα κάνετε ακριβώ από 1η Ιανουαρίου 2012. Εμεί τι να πάμε στι χώρε μα να πούμε στου παραγωγού μα. Αυτού που πληρώνουν το αυξημένο κόστο. Για αυτού τι θα κάνετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλου του συναδέλφου που πήραν το λόγο. Επίτροπε, έχετε το δύσκολο έργο να ικανοποιήσετε όλους τους βουλευτές και να μας καθησυχάσετε για την υλοποίηση αυτών των τόσο σημαντικών μέτρων που εγκρίθηκαν πριν από 12 χρόνια την αίθουσα αυτή κάποιος ως υπουργό συνυπέγραψε για την ε, οδηγία αυτή. Λοιπόν, κύριε Νταλή, το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλες και όλους τους ευρωβουλευτές για, την, ε, για ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ποικίλα ε, σχόλια που θα σας υπόψη σήμερα. Ας προσπαθήσω να δώσω το θέμα στις διαστάσεις του. Εγώ δεν θα μεταφέρω τις ευθύνε μου. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα αρμοδιοτήτων. Ωραία είναι να λέμε τι έκανε η Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι δεν θα, να μην κρατούνται πλέον σε εκλοβούς, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει νομική βάση για να ε, απαγορεύσει την ε, χρήση κλοβών. Είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των χωρών μελών. Εγώ ως Επίτροπος σε διάφορες ε, περιπτώσεις φέτος έθεσα το θέμα υπόψη των χωρών μελών στα ε, Συμβούλια των Υπουργών Γεωργίας, κατ' επανάληψη μάλιστα, για να τους πιέσω να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο της οδηγίας. Εν τέλει όμως είναι δική τους ευθύνη η συμμόρφωση αυτή. Δεν προσπαθώ να πω ότι προς δεν είναι δική μας η ευθύνη. Όλοι μας συνυπάρχουμε σε αυτή την ευθύνη και όλοι πρέπει να αναζητήσουμε μια κοινή λύση. Αλλά επιθυμώ το σώμα σας να κατανοήσει πού ακριβώς έγκυνται οι αρμοδιότητες και ποιοι θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να συμμορφωθούν με τις διάφορες οδηγίες και κανονισμούς που περνούν μέσα από τις νομοθετικές μας διαδικασίες. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι να προσπαθήσω να πιέσω, να οθήσω τις χώρες να δράσουν. Ακόμα και μετά από επανειλημμένες ε, αιτήσει για τη χορήγηση πληροφοριών, ορισμένες χώρες μέλη μέχρι και σήμερα δεν μας έχουν δώσει καν τα δεδομένα της ε, καταστάσεως στη χώρα τους. Η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετωνία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Αυτές λοιπόν είναι οι χώρες οι οποίες μέχρι τώρα δεν μας έχουν δώσει δεδομένα για το που βρίσκεται η κατάσταση στη χώρα τους, στην επικράτειά τους. Έχουμε επίσης το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία που δεν θα συμμορφωθούν πλήρως με την οδηγία. Μετρό λοιπόν 12 χώρες μέλη όπου σημειώνονται προβλήματα. Και δεν λέω ότι όλες οι όρνηθες που ε, εκτρέφονται για την οτοκία σε όλες αυτές τις χώρες αποτελούν το πρόβλημα. Όμως, σε ορισμένες σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό, σε άλλες μικρότερο, της παραγωγής θα είναι παράνομο από την πρώτη Πρώτου 2012. Έχω και το εξή να πω. Στην πολιτική τα θέματα σπανίως έχουν μία και μοναδική διάσταση. Εάν το πρόβλημα ήταν μονοδιάστατο, η λύση θα ήταν εύκολη. Πηγαίνω στους ε, νομομαθείς, οι νομομαθείς μου λένε κάθε αυγό που παράγεται στους κλωβούς αυτούς είναι παράνομο και πρέπει να καταστραφεί. Ωραία λοιπόν. Δέχομαι τότε την πρόταση του κυρίου που μίλησε πριν. Δεν ξέρω πώς. Θα παρέμβουμε. Ωραία, με μια δύναμη, με μια ειδική δύναμη, μια, μια task force από όλες τις χώρες μέλη, να πάμε να καταστρέψουμε όλα τα αυγά, όλους τους κλωβούς, όλες τις όρνηθες που ε, οτοκούν σε αυτούς τους κλωβούς. Αυτή είναι η λύση η προφανής λύση εάν θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα είναι μονοδιάστατο και επιδέχεται μονοδιάστατη λύση. Αλλά το πρόβλημα είναι πολυσχηδές. Έχει και την οικονομική διάσταση στις ίδιες τις χώρες οι οποίες παράγουν τα αυγά. Ορισμένες από τις χώρες αυτές βρίσκονται ήδη σε βαθιά κρίση. Δεύτερον, θα υπάρχει και η διάσταση της επίπτωσης στους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την προσφορά, ζήτηση και βέβαια την τιμή. Άρα θα πρέπει να εξευρεθεί πολιτική λύση. Δεν μπορούμε δηλαδή να αρκεστούμε μονάχα στα νομικά και να πούμε τα αυγά είναι παράνομα, άρα τα καταστρέφουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό που πιέζω εγώ να γίνει και δεν το δήλωσα αυτό διότι ακόμα δεν έχω τη νομική θέση να μπορέσω να το πράξω αυτό είναι να κρατήσω όσα αυγά δεν παράγονται πλέον με την νέα ε, διαδικασία να κρατηθούν τα αυγά αυτά στην ίδια την επικράτεια όπου παράγονται και να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναπαραγωγή και όχι για κατανάλωση. Όμως για την ώρα δεν έχω την απαραίτητη νομική βάση για να επιλέξω τέτοια λύση. Και πιστεύω ότι μια τέτοια λύση ε, θα προστατεύσει τους εκτροφείς και παραγωγούς αυγών που έχουν κάνει επενδύσεις στην χώρα τους ώστε να μην έχουν ανταγωνισμό από φθηνότερα αυγά που έρχονται στη χώρα τους απ' έξω και δεύτερο θα οδηγηθούν όλοι οι εκτροφείς να βελτιώσουν, να διορθώσουν την κατάσταση. Αυτή λοιπόν είναι η λύση που βλέπω. Αλλά δεν μπορώ να σας την υποσχεθώ. Διότι εξακολουθώ να θεωρώ ότι δεν είναι σαφής οι επιπτώσεις. Και εργάζομαι μαζί με τις, με τις υπηρεσίες μου και σε συνεργασία με τις χώρες μέλη για να βρούμε κάποια λύση μέσα στο πλαίσιο αυτό. Αυτά για τις οτό και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πάλι εδώ νομίζω ότι το θέμα των γάμα ταφόμικρων και του μελιού είναι ζήτημα συνύπαρξης πρωτίστως. Άρα, όντως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες συνύπαρξης και ιδίως μεταξύ καλλιεργειών γάμα ταφόμικρων και παραγωγής μελιού και δεύτερον τα σχετικά με τις εγκρίσεις. Και όπως είπα και πριν, Έχουμε ήδη δώσει οδηγίες στην ΕΦΣΑ να αρχίσει την ανάλυση στη βάση της οποίας να μπορούν να χορηγηθούν οι εγκρίσει. Να δούμε δηλαδή πόσο ασφαλής είναι η γύρις μέσα στο μέλι και να μας πούν αν μπορούν να δοθούν εγκρίσει με τον τρόπο αυτό. Και σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια, άκουσα εκεί ορισμένα θέματα που θέσατε, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για τις τροπολογίες αυτές που έχετε καταθέσει όταν θα τις εγκρίνετε, όταν θα τις εγκρίνετε και νομίζω ότι θα είναι μια λύση που μπορεί πράγματι να προχωρήσει θα χρειαστούν κάποιες περαιτέρω συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω ε, εργασία. Ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις ΟΤΟ και θέσεις μου ακόμα και οι Θα απολυθούν ή όχι. Δεν θα πρέπει να παραμείνουν στην πώληση. Αυτή είναι η θέση μου. για να καταλήξουν στον καταναλωτή. Θα είναι περιορισμένο το εμπόριο. Ναι. Θα πρέπει να παραμείνουν δηλαδή στην παραγωγή και όχι να περάσουν στο λιανικό εμπόριο. Βέβαια δεν μπορώ να σας δώσω υποσχέσεις. Αυτό που κάνω είναι να δηλώνω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον προβληματισμό, ποια είναι η προσωπική μου θέση για το θέμα αυτό για την ώρα βεβαίως πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει και μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και με τις χώρες μέλη. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, Σα ευχαριστώ κύριε Ντάλη. Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένοι είναι οι συνάδελφοι με τα απαντήσεις σας. Πάντως σε κάθε περίπτωση το πάθος σου, η ενέργειά σου μας ευχαριστούν ιδιαίτερα. Ε, ίσως σημαντικό είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει ποιος σεβάστηκε τους κανόνες και ποιος όχι. Κάποια λύση θα βρεθεί. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν ξαναζητήσει το λόγο, αλλά δεν μπορώ να τον δώσω σε όλους. Δεν είναι και σωστό. Ένα λεπτό για να χαιρετήσουμε τον Επίτροπο λοιπόν όλο και όλο και μετά θα προχωρήσουμε στο σημείο 6. Grazie. inizio al punto Ευχαριστώ να πάμε στο σημείο 6. Per favore, accomodatevi. Abbiamo solo mezz'ora, poi Έχουμε μόνο μισή ώρα, γιατί μετά πρέπει να συνεδριάσουν οι συντονιστές. 6, Σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Τροποποίηση του κανονισμού 617 του 2009 ΕΚ. Καθίστε παρακαλώ, φτάνει, πρέπει να προχωρήσουμε. Μην κάθεστε όρθιοι στους διαδρόμους, γιατί αλλιώς θα χτυπάμε το σφυρί. Συνάδελφοι, περνάμε στην τροποποίηση του κανονισμού 617-2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομη δασμολογική ποσόστοσης για τις εισαγωγέ βοήου κρέατος υψηλή ποιότητας. Να θυμίσω, συνάδελφοι, πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Λάιον, ότι το θέμα αυτό ανάγεται στο 1998 όταν στο πάνελ διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ κρίθηκε ότι είναι ασύμβατο με τη συμφωνία για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϊγειονομικών μέτρων, η απαγόρευση που είχε εκδώσει η κοινότητα για τις εισαγωγές κρέατος και προϊόντα κρέατος από βοηδή, τα οποία είχαν πάρει αυξητικές ορμόνες. Μετά από μια μεγάλη διένεξη και κυρώσεις που επιβλήθηκαν από ε, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, το 2009 υπεγράφει ένα μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλεπόταν ένας ε, τριπλός μηχανισμός για να μειωθεί το επίπεδο κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη δική της την πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε με τη συμφωνία αυτή να αυξήσει προοδευτικά την ποσόστοση, την δοσμολογική ποσόστοση για τα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας από βοηδή, όπου δεν είχαν, στα οποία δεν είχαν δοθεί αυξητικές ορμόνες ποσόστοση της πρώτης φάσης ορίστηκε σε 20.000 τόνους υψηλής ποιότητας και οριζόταν από τον κανονισμό του Συμβουλίου. Τώρα περνάμε στη δεύτερη φάση, όπως προβλέπει η Συμφωνία με τις ΗΠΑ. Θα πρέπει να ανασταλούν όλες οι αναπομείνασες ε, κυρώσεις κατά της Ένωσης και των προϊόντων της, ενώ από την πλευρά της Ένωσης η αύξηση της ποσόστοσης θα φτάσει τις 25.000 τόνους. Από τους 20 περνάμε στους 45 δηλαδή. Αυτό το θέμα συζητήθηκε και κατά την επίσκεψη στις Ηνωμένε Πολιτείες με τις αρμόδιες αρχές της Αμερικανικής κυβέρνησης και νομίζω ότι σημαντικό είναι να δώσουμε το λόγο ευθύ αμέσως στον Τζόρτζ Λάιον ενώ εποφελούμε τις ευκαιρίες για να χαιρετήσω και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον Διευθυντή Κοτούρνη. Είσαι Κοτούρνη εδώ, ωραία. Έτσι θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για την διοικητική διευθέτηση του θέματος και τις εισαγωγές βόηου κρέατος υψηλής ποιότητας. και δεν θα επικεντρωθούμε μόνο στο τι γίνεται σε κάποιες χώρες. Θα μιλήσει πρώτα λοιπόν ο κύριος Κοτούρνη και μετά ο κύριος Λάιον. Ας δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Κοτούρνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. At, uh, Ήταν πολύ καλή ε, και περιεκτική η εξήγηση που δώσατε για το θέμα αυτό. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω σε αυτά που εξηγήσατε. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω δύο στοιχεία που είναι σημαντικά να τα λάβετε υπόψη. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, οι αναλήψεις που ελήφθησαν από τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ με βάση αυτά τα δύο ξεχωριστά μνημόνια συμφωνίας που συμφωνήθηκαν και υπογράφηκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτές τις δύο συμφωνίες έχουν, ε, οι δύο χώρες συμμορφώθηκαν. Ο Καναδάς ε, ήρε όλες τις ε, κυρώσεις που είχε επιβάλει μέχρι στιγμής και την ίδια άρση ε, φάρμοσαν και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στηρίθηκαν δηλαδή τα μνημόνια συμφωνία και μάλιστα οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, σε σχέση με την 1η Αυγούστου 2012 που ήταν κανονικά η ημερομηνία θέση σε ισχύ της δεύτερης φάσης της συμφωνίας με όλες τις αυξήσεις των εισαγωγών ήδη προκαταβολικά τήρησαν τις συμφωνίες αυτής οι Ηνωμένε Πολιτείε. Επαναλαμβάνω και ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε καλόπιστα εφάρμοσαν τα δύο μνημόνια συμφωνιών. Έχουν άρει όλες τις κυρώσεις και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό συνέβη και 14 μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που ανέφερε την 1η Αυγούστου 2012. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο, ότι οι συμφωνίες αυτές ε, λειτουργούν, ισχύουν και τα αποτελέσματά τους ήταν θετικά. Γιατί είχαμε αρκετά προϊόντα που επηρεάζονταν από τις κυρώσεις ε, και κάλυπταν ενδιαφέραν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχέδιο κανονισμού που έχουμε ενώπιόν μα ε, επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εισέλθει στη δεύτερη φάση και να αυξήσει τι ποσότητε αυτή τη αυτόνομη δασμολογική ποσόστοση και ε, επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις αρμοδιότητες και ε, να αποσύρει ή να αποθηκεύσει ποσότητες αυτής αυτόνομης δεσμολογικής ποσότητας σε περίπτωση που δεν τηρηθούν υποχρεώσεις των εταίρων μας. Μάλιστα, ο κανονισμός ευθυγραμμίζεται με τα οριζόντια θέματα της συνθήκη Λισαβόνα για την επιτροπολογία. Αυτά ήταν τα βασικά ζητήματα της συμφωνίας. Άμεση εφαρμογή λοιπόν των αναλήψεων που ανέλαβαν οι εταίροι μας και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την προβλεπόμενη θέση ισχύ τους. Ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Οπότε θα προχωρήσει η πρόταση και θα εισέλθει στη δεύτερη φάση. Και κατόπιν η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως του χρόνου μπορέσει να προχωρήσει και το επόμενο έτος, το 2013, να καταλήξει οριστική συμφωνία αυτής της διαφοράς με τις ενδιαφερόμενες χώρες και κυρίως με τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοτούρνη. Αν και ε, δεν μου απαντήσατε στη δική μου την απορία, τέλο πάντων ίσω μετά. George Λάιον. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος και Επιτροπή εξήγησαν ποιο είναι το πρόβλημα. Ορμόνες στο βόλιο κρέας. Θα θυμάστε ότι χάσαμε την υπόθεση στο πάνελ του ΠΟΕ σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής ε, βοήου κρέατος που έχει υποστεί ε, επεξεργασία με ορμόνες. Η κάθε άστον προσπαθεί τώρα να ξεπεραστεί ε, το αδιέξοδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείες θα άρουν όλες τις κυρώσεις που ζήτησαν άδεια από τον ΠΟΕ να εφαρμόσουν συμφωνούν να ε, αφήσουν να εγκαταλείψουν τις κυρώσεις και εμείς επιτρέψαμε εισαγωγή ενώ μιας πρώτης ποσόστος 20.000 τόνων και θα φτάσουμε μέχρι τους 45.000 τόνους. Από την άρση των κυρώσεων κερδίζει κυρίως η Ιταλία 99 εκατομμύρια ε, δολάρια ε, αξία, εμπορική αξία Πολωνία, Ελλάδα, Ιρλανδία μαζί με το χείριο κρέας Γερμανία, Δανία, Γαλλία και Ισπανία, Φιλανδία κάτω χώρες, Αυστρία, Βέλγιο, Ρουμανία και Βουλγαρία επίσης, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Πάντως, οι μεγάλοι αποφελούμενοι είναι οι πρώτες χώρες που ανέφερα πριν. Εγώ πρώτα επιθυμώ να ακούσω την συζήτηση που θα διεξαχθεί. Πρόκειται για συναπόφαση. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Για την ώρα δεν προτίθεται να καταθέσω τροπολογίες, αλλά θα κρίνω μετά από την ε, συζήτηση. Είναι απαραίτητο να γίνει σύντομη πρόοδος και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε ε, στις 19-20 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο. Οι ΗΠΑ Πολιτείες ήδη έχουν άρει τις κυρώσεις. Είναι λοιπόν λίγο πιο προχωρημένες από εμάς και ελπίζεται ολόκληρη διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι τον επόμενο Αύγουστο. Είναι σημαντικό θέμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις Ενωμένες Πολιτείες. Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λίγη η διαφορά αποφεύγει την εφαρμογή άλλων κυρώσεων και μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την απαγόρευση εισαγωγής βόηου κρέατος επεξεργασμένου με ορμόνες από τις ΗΠΑ. αν και υπάρχει ένα ποσό κυρώσεων 15 ε, δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων και μετά θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα στη διάρκεια της συζητήσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Τζόρτζ. Και τώρα ο κύριος Λεμπρούν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα συμπληρώνοντα αυτά που ακούσαμε να πω ότι είμαι και σκιώδη για το θέμα στην ομάδα μου. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να χαρακτηρίσουμε το θέμα αυτό ως νίκη ή όχι. Νίκη είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυθεντική ή αν μας εξυπηρετεί τελικά. Μπορεί να είμαστε κάπως ικανοποιημένοι με το διακανονισμό της διαφοράς, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε και κάπως επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Ο τότε επίτροπο Γεωργίας, ο Μισελ Μπαρνιέ, είχε πει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί κατά την θέση εφαρμογή της συμφωνίας και ίσως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης και να εξακριβώσουμε πώς εφαρμόζεται η συμφωνία και να εγγύψουμε και στο θέμα της ποιότητας. Τι εννοούμε βόλιο κρέας καλής ποιότητας, υψηλής ποιότητας. Υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό αυτό μεταξύ των ε, ενδιαφερομένων μερών. Ίσως έτσι αποσπόμαστε κάπως από το βασικό στοιχείο της συζήτησης, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη και η συζήτηση για το θέμα της ποιότητας. Η κυρία Ντελάνς. Μην ανησυχείς, Τζόρτζ, θα είμαι καλή μαζί σου. In Γενικώς, συμφωνώ ότι η κατάσταση εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Ε, όλες τις πλευρές αναφέρατε τις χώρες, αναφέρατε και προϊόντα που ε, δεν, θα τα έβαζαν, έβαζε καν το μυαλό μας, που εν, επλήττονταν από αυτή τη διαφορά την αντιδικία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαιρόμαστε για τη διευθέτησή της. Αλλά ας μην ξεχνούμε και μια άλλη συζήτηση ε, σε ό,τι αφορά τις, τους περιορισμούς για τις παγκόδια κεφαλοπάθεια των βοηθών. Γιατί μιλούμε για το βοηό κρέας, αυξάνουμε την αυτόνομη δεσμολογική ποσόστοση με ε, σε 45-48 τόνους για τις αγωγές βοηού κρέατος. Ε, αλλά θα δούμε πόσο κρέας εμείς ε, πραγματικά εξάγουμε προς τις Πολιτείες. Η απάντηση είναι καθόλου, γιατί οι Πολιτείες δεν έχουν ακόμη άρει τις περιορισμούς τους για τις, ε, για τις παγκόσμια κεφαλοπάθεια των βοηθών, ενώ η Ιαπωνία, ο Καναδάς τις έχουν άρει και αν είμαι καλά ενημερωμένη, η νομοθεσία που θα χρειαζόταν για την άρση των περιορισμών αυτών στις ΗΠΑ ήδη έχει ολοκληρωθεί, έχουν διεκπαιρεωθεί οι έλεγχοι. Το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί η νομοθεσία που ήδη έχει θεσπιστεί. Από ό,τι φαίνεται την περασμένη εβδομάδα έγινε ε, μια επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσως μπορεί να μας το επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετέβη κλιμάκιό της Ηνωμένες Πολιτείες και από ό,τι ακούσαμε γύρω στο 2015 θα αρθούν οριστικά αυτοί οι περιορισμοί που σημαίνει μια ακόμη τετραετία. Γιατί, προς τι, δεν έχουν λόγο αυτοί οι περιορισμοί πια δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω ε, κανονικών τροπολογιών, αλλά νομίζω ότι το σχόλιο είναι εύστοχο, γιατί και τα δύο θέματα, και η αυτόνομη δεσμολογική ποσόστοση και η, η σποκόδηση και κεφαλοπάθεια βοηδών αφορούν το βόηο κρέα. Να ασκήσουμε πίεση στη ΣΥΠΑ, να μην περιμένουμε μια ακόμη τετραετία πριν άρουν του περιορισμού του για την σποκόδηση κεφαλοπάθεια. All Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι πανομοιότυπη με τις προηγούμενες ομιλήτρε. Αυτό εμέσω έχει να κάνει με το θέμα του εξαγόμενου βοήου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Επιτροπή τι έκανε σε σχέση με την άρνηση αυτής τη υπαγόρευση. Ιδίω για την εξαγωγή κρέατος βοηδών, μοσχάρι και βοήου κρέα. Η απαγόρευση υπάρχει ακόμη, ιδίω η καναδική. Είναι τελείω άδικη και έχει να κάνει με το γεγονό ότι 22 κράτη-μέλη έχουν του ίδιου ελέγχου για την κατάσταση σε σχέση με την σπογγόντη κεφαλοπάθεια. Και μάλιστα όπω και στι ΗΠΑ και τον Καναδά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει εμπόριο διατλαντικό μεταξύ Βόρεια Αμερική και αυτών των 22 κρατών. 72 μήνε ε, πέρασε το πρώτο για τους ελέγχους της πογκόντους κεφαλοπάθεια. Και είναι πάρα πολύ μακριά το 2015 για να περιμένουμε να έρθει η απαγόρευση. Έχουμε δείξει όλοι μα την ε, καλή πίστη και την καλή διάθεση. Καιρό να έχουμε και ισότιμου κανόνε παιχνιδιού. Θα έπρεπε λοιπόν η Επιτροπή μα να πιέσει ώστε να βρεθεί μια λύση και σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σμιτ. Ο κύριο Σμιτ. Σύντομο θα είμαι κι εγώ. Συμφωνώ με την φιλοδοξία, με το φιλόδοξο στόχο δηλαδή να υπογραφεί η συμφωνία σύντομα. Βέβαια δεν είμαστε σφραγίδα εδώ της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι και μου φαίνεται λογικό λύθηκε το πρόβλημα των, ορμο, των ορμονούχου βοηδούς να λυθεί το άλλο των μη ρεαλιστικών περιορισμών για την σπουγόδη κεφαλοπάθεια που εξακολουθούν και βρίσκονται σε ισχύ. Λοιπόν, μου φαίνεται λογικό να συνδυαστούν οι προσπάθειες για τις ε, ε ρυθμίσεις των δύο αυτών θεμάτων. Ωραία. Δεν έχουν ζητήσει το λόγο άλλοι. Συνάδελφοι, δεν ξέρω, Τζόρτζ, αν θέλεις να κάνεις κάποια καταληκτικά σχόλια. Γιατί σίγουρα ο κύριος Κοτούρνη κάτι θα θέλει να προσθέσει. Τζόρτζ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έθιξαν αυτό το ζήτημα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά η Επιτροπή αυτή κατά την επισκέψη της στις ΗΠΑ μίλησε με τον Υπουργό Γεωργίας και τον κύριο Κέρτ που είναι πρέσβη επί των εμπορικών θεμάτων και είπαμε και στους δύο ότι θέλουμε να δούμε πρόοδο στα θέματα αυτά. Με τον κύριο Πρόζακ πήγαμε σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Συζητήσαμε λοιπόν τα θέματα αυτά από την πλευρά της Επιτροπής μας και μας είπε ότι μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις πριν το τέλος της χρονιάς. Νομίζω λοιπόν πρέπει την απόφαση αυτή να την ενισχύσουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου αυτού, να ασκήσουμε κάθε πίεση ώστε να αποσπάσουμε περαιτέρω δεσμεύσεις. Τώρα το αν θα υπάρξει τροπολογία για το σχέδιο αυτό έκθεση είναι ανεξάρτητο ζήτημα. Ευχαριστώ να το συζητήσω πάντω με του κοιόδη εισηγητέ και να βρούμε κάποια λύση. Όμω τώρα έχουμε μια ευκαιρία να θίξουμε το ζήτημα και να εντείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ε, προσπάθειέ τη με την αφορμή τη συζήτηση σε αυτό το κοινοβούλιο να αρθούν οι και οι περιορισμοί των ε, σπογκοδο... λόγω τη πογκόδου εγκεφαλοπάθεια. Βέβαια, οι ΗΠΑ ε, ε, έχουν το επιχείρημα ότι τέτοιοι περιορισμοί ισχύουν και για ασιατικέ χώρε. Αλλά καλό θα ήταν να δείξουν συνέπεια οι ΗΠΑ και το ζήτημα να πληθεί για, τις, για την αγορά μοσχαριού, κρέατος μοσχαριού από τις κάτω χώρες, εδώ είναι πολύ σημαντικές οι συνέπειες. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Θέλουμε λοιπόν να είναι η το μήνυμα που θα περάσει από την Επιτροπή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΗΠΑ. Ε, το 2015 είναι πραγματικά πολύ απαράδεκτο μακρινό. Οι σκιώδεις λοιπόν οι εισηγητές και όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν ώστε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και να το προωθήσουμε. Κυρία Λάνη, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Από... Ναι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, θέλει να μιλήσει, αποποιείται τις δευτερολογίες. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Επιβεβαιώνεται ότι στη διάρκεια της επίσκεψης ε, του κ. Νταλή στι ΗΠΑ, του Επιτρόπου Νταλή, αναφέρθηκε το 2015, δηλαδή η άρση ε, περιορισμών μετά από μία τετραετία. Γιατί φαίνεται ότι άλλη εντύπωση αποκόμισαν οι ευρωβουλευτέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το επιβεβαιώσουμε. Αν δεν μπορεί κανεί να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τι πληροφορίε ε, σήμερα, τουλάχιστον να το κάνει γραπτό μέχρι την επόμενη μα συνεδρίαση, γιατί είναι χρήσιμη πληροφορία αυτή. Καλώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Κοτούρνη εκπρόσωπος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρεξήγηση έγινε, δεν αποποιήθηκα ε, τι δευτερολογίε. απλώς περίμενα να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Λάιον. Σε ό,τι αφορά τη σπογγόδια κεφαλοπάθεια βοηδών, ο Επίτροπος ε, Ντάλι έφυγε πριν από λίγα λεπτά τη συνεδρίαση και ήταν στι ΗΠΑ πριν από δύο εβδομάδε και έθιξε αυτό το ζήτημα μεταξύ άλλων με του τέρου μα. Ε, και το ίδιο έγινε και από τον ε, Επίτροπο Τσόλος τέλη Φεβρουαρίου ε, στην Ουάσιγκτον. Και η απάντηση που λάβαμε ήταν παρόμοια με αυτή που μας μετέφερε και ο κύριος Λάιον, ότι η δημοσίευση του, της νομοθεσίας αυτής που είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις από τον κλάδο και τους ενδιαφερόμενους θα ξεκινήσει στα τέλη του έτους. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά και ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης στη διάρκεια του 2012, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, μέσα 2012, δεύτερο εξάμεινο του 2012, στην καλύτερη περίπτωση, θα εγκριθεί το σχετικό νομοθέτημα. Δεν νομίζω ότι το 2015 είναι διορία που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όντω ε, εύστοχα τα σχόλια για την σποκώδη κεφαλοπάθεια, παρόλο που δεν είναι θέμα άρρητα συνδεδεμένο με το μνημόνιο συμφωνία. αλλά σίγουρα υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε κλείνουν τις πόρτες στις εισαγωγέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα ζητούν από την Κορέα και την Ιαπωνία να επιτρέψουν τα δικά του προϊόντα στι δικέ του αγορές παρά το δικό του εσωτερικό πρόβλημα σποκόδου εγκεφαλοπάθεια. Θα πρέπει να είναι συνεπή. Υπάρχει πίεση πάντω προ τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πολλοί παραγωγοί έστειλαν επιστολέ στον αρμόδιο υπουργό και στον κύριο Κίρκ ζητώντα διευθέτηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και εσωτερικά λοιπόν μεγάλη πίεση και πιστεύω ότι η πολιτική βούληση θα ακολουθήσει και θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις του Ηνωμένες Πολιτείες και θα δημοσιεύσουν μέχρι το τέλη του έτους την πρόταση. Πάντως και οι δύο επίτροποι και ο κύριος Ντάλη και ο κύριος Τσόλος έθιξαν αυτό το ζήτημα στις επαφέ τους με τους ομολόγους της Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, κάτι που παρέλειψα από την πρώτη μου εισαγωγή, ε, την ερώτηση του κυρίου Κάστρο, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη αυτόνομη δασμολογική ποσότητα. Αυτό αφορά ένα τμήμα των εισαγωγιών, όχι όλου. Υπάρχει πίεση ώστε να μιληθούν όσο το δυνατόν περισσότερε άδειε και υπάρχει πληθώρα αιτήσεων για αυτόνομη δασμολογική ποσότητα, κάτι που δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον και που οδηγεί σε μικρή κατανομή των αδειών μεταξύ των εισαγωγιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, άλλαξε τη διοίκηση πριν ε, τα, τα, τις διοικητικές διατυπώσεις πριν α, τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά μάλλον ήταν απο, αναποτελεσματικά τα μέτρα. Είχαμε ευρύτατες διαβουλεύσεις με τον κλάδο και τους εισαγωγείς και οι α, Αμερικανοί εξαγωγεί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και μαζί του είχαμε συνομιλίε. Και τώρα προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι ο καταλληλότερο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που δημιουργεί εκνευρισμό και ανησυχίε, τουλάχιστον σε ένα τμήμα των εισαγωγέων η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας γνωστοποιήσει τη θέση της. Πάντως είναι ίσως ένα θέμα που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του TRQ. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως στο μέλλον δημιουργηθεί μια κλιμάκωση και ασκηθεί περαιτεροποίηση. Αυτή τη στιγμή, παραλαμβάνω, δεν επηρεάζει την εφαρμογή του TRQ, της αυτόνομης θεσμολογικής ποσόστοσης γιατί οι ροές εισαγωγών-εξαγωγών είναι απρόσκοπτες μέχρι στιγμής. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Ε, Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον δόκτωρα Κοτούρνη για την απάντηση που μας έδωσε. Είναι σημαντικό όσο περισσότερα κράτη γίνεται να συμμετάσχουν και να μην περιοριστεί όλο αυτό σε ορισμένους μόνον. Νομίζω ολοκληρώσαμε τα σημεία μας. Ένα λεπτάκι διάλειμμα και συνεχίζουμε με τις συνεδρίες των συντονιστών. Η Επιτροπή μας συνεχίζει κανονικά αύριο το πρωί στις 9. Ευχαριστώ όλους. Συντονιστές, παρακαλώ, παραμείνετε στην αίθουσα. Θα αρχίσουμε αμέσως.